Good morning everybody. Apologies that I couldn't be with you yesterday. Καλή σας μέρα. Συγγνώμη που δεν ήμουν μαζί σας χτες για προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους διεύθυναν την Επιτροπή. Ε, η, το κομμάτι για την, τον εντελεχή νομοθετικό έλεγχο θα καλύψει σήμερα την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών. Στο τέλος αυτού του κομματιού πριν την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα σας ενημερώσω για τον τριμερή διάλογο για την, ε, ε, για την ηλεκτρονική ψηφιακή, για την ψηφιακή αγορά τηλεπικοινωνιών. Schreiber. Ο κ. Σράιμπερ είναι εδώ από κοινό Κομισιόν, ε, διευθυντής για το ΚΟΣΜΕ, από τη Γενική Διεύθυνση ε, Εσωτερικής ε, Αγοράς, Μικρομισιών Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας. Θα μας ενημερώσει για την εφαρμογή της οδηγίας καθυστερήσεων πληρωμών. Θα μπορούσατε να ξεκινήσετε ενημερώνοντάς μας για το πού βρισκόμαστε και μετά θα ακούσουμε τις ερωτήσεις των μελών που ενδιαφέρονται. Thank you, and good morning, everyone. Um, Καλή σας μέρα. Χαίρομαι που είμαι ξανά μαζί σας. Από 1η Ιουνίου έχω αλλάξει καθήκοντα, ε, οπότε ζητώ ε, ε, να με αντιμετωπίσετε με ε, κατανόηση γιατί είμαι καινούργια, έχω και τον κύριο Αντρόπουλο δίπλα μου ε, που θα μας βοηθήσει επίσης. Θα σας μιλήσω για την ε, σωστή εφαρμογή της οδηγίας καθυστερήσεων πληρωμών. Οι πληρωμές και οι εμπορικές ανταλλαγές ανάμεσα στις οικονομικές φορείς και ανάμεσα στις οικονομικές φορείς και ε, δημόσιες αρχές, ε, κρατικές αρχές είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες προθεσμίες. Οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν πολύ αρνητικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και περιπλέκουν την διαχείρισή τους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και εμπίπτουν στις δικές μας αρμοδιότητες, στις αρμοδιότητες της γενικής μας διεύθυνσης οι πολλές οδηγίες επηρεάζουν την ζωή των μικροσύνων επιχειρήσεων, όμως ιδιαίτερα αυτή ακριβώς η οδηγία, ιδιαίτερα στο δεδομένο περιβάλλον κρίση το οποίο ζούμε. Γνωρίζετε την οδηγία νομίζω, αλλά να σας ενημερώσω για το ποια είναι τα τέσσερα βασικά της χαρακτηριστικά, οι τέσσερι βασικές της διατάξεις. Η εναρμόνιση της περίοδου πληρωμών από τις κρατικές αρχές προς τις επιχειρήσεις καταρχήν. Ε, εδώ έχουμε μια προθεσμία 30 ημερών. Με πολύ λίγες εξαιρέσεις. Μετά έχουμε την ελευθερία ε, σύναψη συμβάσεων ε, και την χρονική προθεσμία 60 ημερών για πληρωμή εκ μέρους των επιχειρήσεων, από επιχείρηση. Μετά έχουμε ε, αυτόματη εφαρμογή του δικαιώματος εισπραξής ε, ε, τόκων υπερημερίας. Και τέλος, ε, το, το επιτόκιο αυτό καθορίζεται από τον νόμο στο 8% επιπλέον ε, του βασικού επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας. Να σας πω που βρισκόμαστε. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν ενημερώσει την Κομισιόν, έχουν κοινοποιήσει την Κομισιόν τον Ιούλιο του 2014 το τελευταίο για την μεταγραφή της οδηγίας και από ό,τι φαίνεται οι περισσότερες μεταγραφές έχουν γίνει σωστά με ελάχιστες εξαιρέσεις τις οποίες παρακολουθούμε προσεκτικά από πλευρά της Κομισιόν. Έχουμε μάλιστα ξεκινήσει και τρεις διαδικασίες επί παραβάση για κακή μεταγραφή ε, της οδηγίας. Ε, και αυτές όμως ε, πιθανότατα θα επιλθούν σύντομα. Το πιο σημαντικό είναι όμως ε, το κατά πόσον, εφαρμόζεται σωστά η οδηγία ε, ανεξάρτητα από το αν έχει μεταγραφεί σωστά ή όχι. Έχουμε ξεκινήσει ε, διαδικασία υπερβάση για κακή εφαρμογή της οδηγίας εναντίον τριών χωρών Ισπανίας, Ελλάδας και Ιταλίας. Οι καθυστερημένες πληρωμές από πλευράς των κρατικών αρχών σε αυτές τις χώρες είναι ένα γνωστό φαινόμενο, επιβεβαιώθηκε άλλωστε από τα πολλά παράπονα ε, που λάβαμε. Ε, προκειμένου να αξιολογήσουμε το αν εφαρμόζεται σωστά η, η οδηγία αυτή σε άλλες ε, χώρες, η Γενική Διεύθυνση Grow ξεκίνησε μια μελέτη, κάτι το οποίο κάνουμε συχνά άλλωστε και με άλλες οδηγίες, σε αυτή τη ε, μελέτη θα αξιολογήσουμε τις πρώτε, τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής της οδηγίας στα 28 κράτη-μέλη και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα συμπεριληφθούν στην έκθεσή μας μαζί με άλλα πορίσματα που θα έχουμε, έκθεση που θα υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το Μάρτιο του 2016, κάτι που προβλέπεται έτσι κι αλλιώς από την οδηγία. Όλα αυτά ως μια γενική επισκόπηση της ε, κατάστασης ε, αυτή τη στιγμή. Ε, βασιζόμαστε πολύ σε καταγγελίες που λαμβάνουμε, αλλά ταυτόχρονα παρακολουθούμε και τις, ε, και τις πληροφορίες που βρίσκονται ε, δημοσιευμένες, οποιασδήποτε πληροφορίες ή νούμερα βλέπουμε δημοσίως, τα λαμβάνουμε υπόψη. Αυτά είναι η γενική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε και ερωτήσεις. Να σας ε, συνοψίσω όμως ότι η κατάσταση είναι αρκετά ικανοποιητική σε ό,τι αφορά την πραγματική ε, μεταγραφή της οδηγίας. Όμως δεν είναι εξίσου ικανοποιητική σε ορισμένα κράτη-μέλη τουλάχιστον ε, σε ό,τι αφορά την σωστή εφαρμογή της. Thank you very much for that. Ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλετε να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις, να ακούσουμε ένα πρώτο κύριο ερωτήσεων και μετά να επανέλθουμε. Και ξεκινάμε με ε, τον κύριο Στεφανίτσε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Σράιμπερ για την παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης. Το επίπεδο αυτό, αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για τους οφειλέτες και για τις πληρωμές σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχουν περισσότερα ε, προγράμματα όσον αφορά αυτή την οδηγία. Έχω δύο ερωτήσει. Η πρώτη αφορά τη μαύρη λίστα ε, των οφειλετών. Ε, έχετε κάποια τέτοια εμπειρία με τις μαύρε λίστες οφειλετών που ενδεχομένω δημιουργούνται κατά χώρα. Υπάρχουν κάποια κράτη μέλη που έχουν κάποιε καλύτερε πρακτικέ στην κατάρτιση τέτοιων μαύρων λιστών ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, γιατί ξέρετε επικεντρωνόμαστε στις ε, καθυστερήσεις πληρωμών μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και στις καθυστερήσεις κρατικών πληρωμών αλλά το μείζον ζήτημα αφορά την ε, συμμετοχή των κρατών μελών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Σκοπεύετε λοιπόν να συμπεριλάβετε και αυτές τις συμμετοχές των κρατών μελών στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οδηγία αυτή για την καθυστέρηση πληρωμών, ευχαριστώ στον Νίκολα Ντάντη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που έχουμε σήμερα το πρωί να εξετάσουμε αυτή την πολύ σημαντική οδηγία που θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα της εσωτερικής αγοράς μέσω κανόνων τέτοιων που θα επιτρέψουν σωστές οικονομικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων μεταξύ τους και μεταξύ επιχειρήσεων και κρατικών μηχανισμών. Εγώ, η δική μου χώρα βρίσκεται στη μαύρη λίστα. Έχει συσσωρεύσει μέσα στα χρόνια από τα υψηλότερα χρέη του κρατικού, του κρατικού μηχανισμού. Πολύ ψηλό χρέος. Το έχουμε δει και είναι ένα από τα θέματα που έχουν επιχειρήσει να αντιμετωπίσουν οι τελευταίες κυβερνήσεις στη χώρα μου ε, όχι μόνο για να ανταποκριθούμε στη διαδικασία παραβάση που έχει ξεκινήσει από την Κομισιόν ενώπιον της Ιταλίας, αλλά και για να καταστήσουμε πιο αποτελεσματικό το οικονομικό σύστημα και να εξαλείψουμε αυτή τη δομή της αγοράς. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρχει αυτό το θέμα υπό εξέταση και που η Κομισιόν παρακολουθεί σταθερά την εφαρμογή της οδηγίας. Στο τελευταίο κομμάτι είπατε ότι είστε ικανοποιημένοι από τη μεταφορά της οδηγίας αλλά λιγότερο από την εφαρμογή και από τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί. Εμείς θα θέλαμε να βελτιωθούν και αυτά τα αποτελέσματα και η εφαρμογή. Εμείς θέλουμε να σας ρωτήσουμε στη διαδικασία αυτή παρακολούθησης προσπαθείτε να παρακολουθήσετε και τις βέλτιστες πρακτικές βελτιστές πρακτικές που εφαρμόζονται σε ορισμένες χώρες ε, μέσω εναλλακτικών λύσεων ε, για την επιτάχυνση της, ε, των καθυστερημένων πληρωμών οι οποίες έχοντας σωρευτεί μέσα σε πολλά χρόνια δημιουργούν ελαττώματα και προβλήματα στη δημόσια οικονομικά τα οποία μετά έχουν επιπτώσεις γενικότερα στις χώρες και στα ευρωπαϊκά οικονομικά. Στην ανάλυση λοιπόν αυτή που κάνατε Έχετε κάποιο ε, ε, λίστα βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη για να ανταποκριθούν στι απαιτήσει και στους στόχους της οδηγίας. Ευχαριστώ, Ντίτερ Σάνζελ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση. Περιμένουμε βεβαίω την έκθεση αξιολόγησης που θα κατατεθεί του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε κάποιες ιδέες για το πώς θα διατυπωθεί αυτή. Ε, προετοιμαζόμενοι για τη σημερινή συζήτηση, ε, ρώτησα γύρω μου πληροφορίες για το πώς αποδίδει αυτή η οδηγία. Από τον χώρο των επιχειρήσεων οι απαντάσεις ήταν είτε χαρακτηριστικά αρνητικές είτε ε, απόλυτης άγνοιας και από την ε, ιδιαίτερη μου πατρίδα μαθαίνω ότι μπορεί να εφαρμόζεται μένα αλλά δεν ξέρουν αν λειτουργεί. Η ε, νομοθεσία δεν επιβάλλει στα κράτη-μέλη να παρακολουθούν την υλοποίηση της οδηγίας και έτσι δεν είναι γνωστό καν αν υπάρχουν τα σχετικά δεδομένα. Γι' αυτό νομίζω ότι ήταν λάθος ο τρόπος της μεταφοράς και ανησυχώ βλέποντας ότι στο σύστημα μεθοδολογίας που τη διαφάνειά σας, στο σύστημα και τη μεθοδολογία που τη διαφάνειά σας, αναφέρεστε σε επιστημονική προσέγγιση. Εγώ θα ήθελα οι εμπλεκόμενοι φορείς να δίνουν την αξιολόγηση και μάλιστα και με συνεντεύξεις οι οποίες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές για να καταλάβουμε καλύτερα εάν λειτουργεί στην πράξη η οδηγία αυτή. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρει αυτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσει δεν πρόκειται να κάτσουν να ασχοληθούν με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων σας. Και ελπίζω να μπορέσετε να ασχοληθείτε και με τις θέσεις των ε, εμπλεκομένων σε όλα τα κράτη-μέλη. Το τουλεχθέντο έχω μια ερώτηση. Διευθύντρια. Πώ μπορείτε να εξασφαλίσετε και εάν να εξασφαλίσετε ότι ενημερώνονται πλήρω οι μικρομεσαίε επιχειρήσει για τα δικαιώματά τους, για το πεδίο και το αντικείμενο της οδηγίας, ε, για το ότι ενδεχομένω ε, ε, έχουν αξίωση για αποζημίωση. Ένα από τα αίτια που παρουσιάζονται ως προς την μη υλοποίηση και με γνώση από τις επιχειρήσεις της ε, ύπαρξης αυτής της ε, οδηγίας, όσο περιστασιακά και αν είναι αυτά, δείχνουν ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Κάνω λάθος και τι μπορούμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δίο. Δε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και για την ευκαιρία ιδιαίτερος που μας δόθηκε να συζητήσουμε την οδηγία αυτή. Ήταν μία από τις πρώτες που συνάντησα ως ε, βουλευτή στην προηγούμενη θητεία στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Όπως είπε και η Ντίτα, έχει ζωτική σημασία για τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και είναι απαραίτητο να λειτουργήσει σωστά. Και όπως είπαμε, η επιστημονική προσέγγιση δεν ε, είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να ασχοληθώ με το θέμα αυτό. Είχαμε διάφορα ζητήματα για την, ε, που είδαμε στη συζήτηση για την οδηγία και που έχουν να κάνουν με την ε, εξουσία. Με ποια έννοια, ότι όταν μια μικρομεσαία επιχείρηση έχει συνάψει σύμβαση, η οποία δεν λειτουργεί ικανοποιητικά με, την, με τις τοπικές αρχές, ε, δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί εύκολα γιατί προσβλέπει σε μια περαιτέρω σύμβαση και θα χάσει αυτή την ευκαιρία. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε λοιπόν. Και βέβαια στην έκθεση τη Επιτροπή πρέπει να καταγράφεται. Και με ενδιαφέρει περισσότερο όχι τόσο η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο όσο η διάρθρωση της οδηγίας, η δομή της μέσα στο εσωτερικό πολιτιακό πλαίσιο για την ε, κάλυψη αυτού του προβλήματος των καθυστερημένων πληρωμών. Επίσης, η ισότητα των όπλων είναι πολύ δύσκολο για τις μικρές επιχειρήσεις να στραφούν δικαστικά εναντίον μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Είπαμε ότι υπάρχει ένα διάστημα κατά το μέγιστο 60 ημερών. Ναι, αλλά μια μικρή επιχείρηση δεν θα αισθανθεί ασφαλής ότι θα υλοποιηθεί η οδηγία σωστά. Και ρωτώ, κράτη-μέλη, τα οποία ενδεχομένως έχουν και εταιρείε δημοσίου που ανήκουν στο δημόσιο, θα επιτρέπουν με τις διατάξεις στις μικρότερες επιχειρήσεις να σταθούν στο πλαίσιο αυτή της οδηγίας. Και θυμάμαι ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε τόσο καλέ επιδόσει, τουλάχιστον στο παρελθόν, όταν είχαμε μελετήσει την υπόθεση. Είχαμε δει προβλήματα προ τι καθυστερήσει, τι πληρωμέ, που διαπιστώνουμε ακόμη και με το, η διαδικασία του προπολογισμού. Η Επιτροπή έχει κάποια πιο πρόσφατη αξιολόγηση των δικών της επιδόσεων ως προς τις ε, καθυστερημένες πληρωμές. Η Πρόεδρος. Ακούω ε, από την κάθε ομάδα, ανάλογα με τον ποιον έχει ορίσει η ομάδα ως εκπρόσωπο στη συζήτηση αυτή, κυρία Γκραπίνη, για να ε, τις ακούσουμε με τη σειρά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, και θα ήθελα να πω ότι το θέμα αυτό εγώ το συνάντησα πριν ασχοληθώ με την πολιτική. Ε, όταν εργαζόμουν σε μικρομεσαία επιχείρηση και ιδιαίτερως με ενδιαφέρει αυτή η οδηγία, έχω συμμετάσχει και σε συζητήσει στη Ρουμανία. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξή. Η οδηγία είναι βέβαια καλή ως ιδέα. Υπάρχει όμω ένα πρόβλημα και το θίγω εδώ. Το έχω άλλωστε θίξει και στο παρελθόν. Η θέση εφαρμογή τη οδηγία κατέλαβε να εξαπίνει στα κράτη-μέλη, γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πολύ διαφορετική ανάλογα με το κάθε κράτο. Προπολογισμό των επιχειρήσεων που ενδεχομένω παρουσιάζουν σημαντικέ καθυστερήσει στι πληρωμέ, μεγάλε επιχειρήσει σε σχέση με το κράτο ή μικρέ επιχειρήσει σε σχέση με μεγάλε επιχειρήσει. Και προσπάθησε η Ρουμανία να ε, καταρτήσει έναν ε, πίνακα, μια μαύρη λίστα θα λέγαμε, εκείνων των επιχειρήσεων που δεν είχαν εξοφλήσει του προμηθευτέ του. Η Επιτροπή όμως μας κάλεσε να σταματήσουμε την πρωτοβουλία αυτή. Μπορεί να αναφέρονται 60 μέρες στην οδηγία, αλλά μας λέτε ότι αυτό ε, αφορά τη σχέση μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων εφόσον δεν προβλέπεται κάτι αντίθετο στην ε, συμβατική σχέση, στην ε, σύμβαση. Ε, ναι, αλλά μια μικρή επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τους όρους μιας σύμβασης. Για τα 40 ευρώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν τα εισπράττουν. Τι θα κάνουν λοιπόν, πώς θα μπορέσουν να στραφούν κατά μίας ε, μεγάλης επιχείρησης για να διεκδικήσουν την, ε, το καταποκοπήν αυτό ποσό. Σε πολλές χώρες, άλλωστε και στη Ρουμανία που γνωρίζω καλύτερα, δεν υπάρχουν ε, εμποροδικεία. Άρα δεν είναι εύκολες οι διαδικασίες για να προσφύγουν οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι πιο αδύναμες οικονομικά. Έχετε κάποιο μηχανισμό για να εξασφαλίσει τη λειτουργία του συστήματος σε εθνικό, σύστημα, σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να μην χρειαστεί να πέρασε από ένα μακρύ και βαρικίνητο σύστημα ε, δικαστικό η επιχείρηση. Και επίσης θα ήθελα μια διευκρίνηση ως προς το κατά πόσον χωρεί βελτίωση αυτής της οδηγίας. Όταν πρόκειται για καθυστερήσεις ε, πληρωμών από αρχές τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, και αν υπάρχουν μέτρα που μπορούμε να εισαγάγουμε έτσι ώστε να επιλύονται οι διαφορές όχι με μία μακρά και βραδικίνητη διαδικασία δικαστική, αλλά με άλλες πιο ευκίνητες διαδικασίες για να διευκολυνθεί και η μικρομεσαία επιχείρηση και να μην χρειάζονται χρόνια για να ανακτήσει τα μη καταβληθέντα ποσά. Μπορεί να δίνετε εντύπωση ότι έχει μεταφερθεί σε εθνικό επίπεδο η οδηγία, αλλά εάν κάνετε τη μελέτη τη πραγματική υλοποίηση και των συστημάτων που λειτουργούν, θα δείτε ότι δεν έχει επιτευχθεί είτε η ίσπραξη είτε των μη καταληφθέντων ποσών είτε των τόκων υπερημερία ε, με βάση την οδηγία αυτή. Η πρόεδρο. Εφόσον δεν θέλει κανεί άλλο το λόγο, να σα πω εγώ ποια είναι η άποψή μου. Ε, ήμουν και ηγητή την εποχή που εγκρίναμε αυτή την ε, οδηγία. Ε, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο κ. De Young, ε, De σε ό,τι αφορά την απόδοση και την επίδοση της Κομισιόν ε, που δεν ήταν και πολύ καλή σε εκείνη τη φάση. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό να το δούμε γιατί πρέπει και εμείς να δίνουμε το καλό παραδείγμα. Αλλά ε, να πω για το όσα είπε η κυρία Τσαραντζόβα σε ό,τι αφορά τις συμβουλές που μπορούμε να δώσουμε προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, τι συμβουλέ θα μπορούσαμε να δώσουμε σε ό,τι αφορά την ερμηνεία ε, του, του όρου ε, καταφανώς άδικο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να θα πρέπει να μπορούν να διαπραγματεύονται μακρύτερες ε, περιόδους, ε, παράδειγμα ε, ο κλάδος των, των κατασκευαστικών προϊόντων ή των μαγαζιών που πουλούν προϊόντα μαστορέματος, do it yourself, και ήθελα να δω αν αυτές οι μακρύτερες περίοδοι που είναι απαραίτητε για αυτούς τους κλάδους θεωρούνται καταφανώς άδικες ε, ή πώς τις, ε, έχει χειριστεί, ε, έχουν χειριστεί τα κράτη-μέλη αν μπορούμε δηλαδή, αν η οδηγία δίνει ευελιξία την οποία όμως κάποιοι ενδεχομένως καταχρώνται ή όχι. Η κυρία Γκέπχαρτ και ο κύριος Φαπ παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πολλέ από αυτέ τι ερωτήσει θέλω και εγώ να διατυπώσω. Δεν θα τι επαναλάβω λοιπόν. Θα σταθώ σε ένα σημείο το οποίο μα είχε απασχολήσει και όταν κάναμε το νομοθετικό έργο. Ιδιαίτερα. Δυστυχώ δεν έχω προχείρω το κείμενο. Αλλά δεν γνωρίζω κιόλα τι είχε αποφασιστεί ω προ τον ορισμό του δημοσίου Ερωτώ λοιπόν τη δημόσια αρχή. εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νοείται ω Δημόσια Αρχή και αν τηρεί αυτή την οδηγία. Ευχαριστούμε. Ο Ανδρέας Σουά, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι στου ορισμού πρέπει να κάνουμε μια διάκριση στην οδηγία για την καθυστέρηση πληρωμών, ότι μπορεί να υπάρχει μια ομάδα κρατών η οποία παρά την ε, πάροδο τη ε, περίοδου μεταφορά δεν την έχει μεταφέρει σε εθνικό δίκαιο και άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί ουσιαστικά το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γι' αυτό έχω να κάνω μια ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα προ την κυρία Στάιμπερ. Ποιοι είναι οι λόγοι για του οποίου τα κράτη αυτά δεν έχουν μεταφέρει σε εθνικό δίκαιο, είναι αδυναμία δημοσιονομική, δεν εμπόρεσαν να τηρήσουν τι προθεσμίε για λόγου ε, οικονομικού, δηλαδή το ξέχασαν, ε, υπάρχει τρόπο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν είχε γίνει η συζήτηση γενικά για την ε, διακυβέρνηση ότι οι διαδικασίες επί παραβάση Όπω είχε πει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν διευκολύνουν πάντα, δεν δίνουν λύση στα προβλήματα και είχε πει η Επιτροπή δεν βοηθούν, πρέπει να πείθουμε τα κράτη να μεταφέρουν τι οδηγίε. Άρα αυτό θα πρέπει να μα βάλει σε σκέψει για την υλοποίηση τώρα. Καλό είναι μαζί με τα ξερά να μην καίμε και τα χλώρα. Γιατί έχουμε να κάνουμε με μια ρύθμιση η οποία έπρεπε να εσωματωθεί στο εθνικό αστικό δίκαιο. Άρα, ναι, μεν είναι πολύ καλό να το γνωρίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά από την άλλη έχουμε πολύ περιορισμένες δυνατότητες να ε, προβάλλουμε, ε, να διαφημίσουμε με αυτή την έννοια το εθνικό αστικό δίκαιο γιατί είναι διαφορετικό στα 28 κράτη-μέλη. Είναι κάτι διαφορετικό από το να βάλουμε σε ένα αεροδρόμιο μια πινακίδα που θα λέει να ξέρετε ποια είναι τα δικαιώματά σου σε επιβάτη. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό με το αστικό δίκαιο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει κάθε κράτο να κάνει την προσπάθειά του ή διαφορετικά να φτάσει μέχρι τα δικαστήρια και να πάρει την, ε, ε, την απόφαση για τη συγκεκριμένη υπόθεση κάθε δικαστή όταν έρχεται η ώρα. Η πρόεδρο, πολλέ ερωτήσει. Εάν έχει την καλοσύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τι απαντήσει. και ίσως αν έχετε την καλοσύνη να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για τις εκρεμείς δίκες επί παραβάση. Σε ποιους τομείς αναφέρονται. Yes, thanks. Let me run through the... Λοιπόν, να απαντήσω τις ερωτήσεις, ξεκινώντας από την κυρία Στέφανης και την Αυρελίστα. Φυσικά έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τις μαύρες λίστες σε διάφορους τομείς, αλλά σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, δεν θα ήταν το καταλληλότερο εργαλείο, διότι το ζήτημα αφορά κυρίως καθυστέρηση πληρωμών από δημόσιε αρχές. Εστιάζεται περισσότερο σε αυτά τα προβλήματα. Οπότε μην νομίζετε ότι θα χρειαζόμαστε μια μαύρη λίστα εμπορικών επιχειρήσεων, διότι το πρόβλημα είναι κυρίως οι κρατικές αρχές, οπότε Καλό θα ήταν ε, αφού έχουμε ε, ε, προβλήματα στην Ιταλία, στην Ισπανία κτλ. Υπάρχει τεράστια πίεση προς τις δημοσιαρχές, οπότε η μαύρη λίστα θα ήταν ένα μέσο το οποίο θα ήταν αναποτελεσματικό σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο. Ευχαριστούμε για την ευαισθητοποίηση που αναφέρατε ότι πρέπει να έχουμε και ε, θα ακούσετε ουσιαστικά επιχειρήσεις που θα σας αναφέρουν ζητήματα οπότε είναι σημαντικά να μαθαίνουμε τέτοια σχόλια από τις επιχειρήσεις ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε σωστά κατά πόσο νομοθεσία μας εφαρμόζεται σωστά επί τόπου ή όχι. Για την κυρία Τσαράζοβα Αυτό που λέτε ότι η οδηγία δεν απαιτεί από τα κράτη-μέλη να παρακολουθούν την εφαρμογή δεν είναι απόλυτα σωστό. Τα κράτη-μέλη όμως ε, υποχρεούνται να μεριμνούν για τη διαφάνεια, για την ευαισθητοποίηση, υπάρχει το άρθρο Υπάρχει λοιπόν κάποια υποχρέωση προς τα κράτη-μέλη να μεριμνούν και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή της οδηγίας παρότι εντάξει, δεν χρειάζεται να συντάξουν κάποια έκθεση αλλά είναι σαφές ότι έχουν και την υποχρέωση να παρακολουθούν ότι λειτουργεί αποτελεσματικά και η οδηγία τώρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς έχουμε κάνει διάφορες ενημερωτικές εκστρατείες σε όλα τα κράτη-μέλη για την ενημερωσή τους και στην Τσεχική Δημοκρατία όπου συγκεντρώνουμε δημόσιες αρχές ε, ενώσεις επιχειρήσεων και φυσικά έχουμε και τα ευρωπαϊκά δίκτυα και άλλα ενημερωτικά δίκτυα που φέρνουν αυτές, μεταφέρουν αυτές τις πληροφορίες ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φυσικά πάντα υπάρχουν και περισσότερα που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά έχει γίνει κάποια εκστρατεία στοχευμένη, ενημερωτική. Για τον κύριο Ντεγιόγκ, και άλλους που έθεσαν το ίδιο ζήτημα τι γίνεται για την Επιτροπή και φανταζόμαι και για το Κοινοβούλιο σε αυτού του. Και εμείς είμαστε κριτικοί οργανισμοί, οπότε η οδηγία ισχύει και για μας. Δυστυχώς δεν έχω ακριβή νούμερα αυτή τη στιγμή. Αλλά από όσα μου είπαν, γιατί ήταν η πρώτη ερώτηση που έκανα και εγώ όταν ανέλαβα αυτή την εργασία, είπα και εγώ αποτελούμε υπόδειγμα. Ε, υπάρχει μια κατάσταση που θυμάμαι από πριν μερικά χρόνια. Ε, η κατάσταση παλιότερα ήταν, δεν ήταν πολύ ικανοποιητική, αλλά νομίζω τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα, αλλά ναι, σίγουρα ισχύει αυτό και για τα δύο όργανα, την Κομισιόν και εσά. Και πρέπει να αποτελούμε υπόδειγμα το ζήτημα που ανέφερε ο κ. Δεγιόν για το πώ μικρότερε επιχειρήσει μπορούν να καταγγείλουν μεγαλύτερε. Ε, αυτό σχετίζεται και με την ερώτησή σας Βίκη για την ερμηνεία ε, ε, υπερβολικά άδικων όρων. Ε, αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορεί να υπάρχει σε οποιοδήποτε τομέα όπου νομοθετούμε. Όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά ε, ισχύως μεταξύ, δύναμης μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Όταν ε, πηγαίνει κανείς και καταγγέλει ένα μεγαλύτερο οικονομικό εταίρο, υπάρχει κίνδυνος φυσικά, αυτό είναι προβληματικό, αλλά είναι δύσκολο να το λύσουμε προσθέτοντας ε, άλλο ένα επίπεδο στην νομοθεσία. Ε, απλά είναι γνωστό ότι αν κάποιος δεν συμμορφώνεται με την οδηγία, αυτό θα γίνει γνωστό. Εάν κάποια επιχείρηση δηλαδή κατά επανάληψη ε, επεκτείνει τις ε, προθεσμίες, παρατείνει τις προθεσμίες, ε, θα γίνει γνωστό. Έχουμε το δίκτυο Enterprise Europe και άλλα όπου μπορούν να ζητήσουν βοήθεια επιχειρήσεις. Δεν ξέρω ποιο το σχολίασε, αλλά ναι, ναι είχατε, ναι, δίκιο. Ένα πράγμα είναι να προσφύγει στο δικαστήριο, αλλά συχνά αυτό δεν βοηθάει μια επιχείρηση από πρακτική άποψη. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορεί να επιληθεί το ζήτημα μέσω της νομοθεσίας αυτής καθεαυτής, αλλά ε, όπως είπα υπάρχουν όλοι αυτοί οι οργανισμοί στους οποίους μπορούν να στραφούν οι επιχειρήσεις για να λάβουν βοήθεια με άτυπο τρόπο ώστε να επιλύσουν μερικές φορές τα ζητήματα εξωδικαστικά να αποφύγουν να πάνε στα δικαστήρια. Αυτή η υποστήριξη και όλοι αυτοί οι σχετικοί μηχανισμοί είναι πολύ σημαντικοί. Ε, τώρα να επανέλθω στην ερώτησή για την Κομισιόν, Αντρέα Φαμπ. Γιατί δεν γίνεται. Α, να συνεχίσω στα αγγλικά, να μην σας κουράζω με τα ακουστικά. Δεν είναι σωστό νομίζω 100% το πρόβλημα, ότι υπάρχει πρόβλημα στη μεταφορά. Είχαμε αρκετά καλό επίπεδο μεταφορά στην αρχή, σχεδόν όλα τα κράτη. Η Ιρλανδία νομίζω που έχει μια δημόσια διαβούλευση εκκρεμή. Ε, θα συμπληρώσει τον αριθμό των κρατών μελών που έχουν μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Το πραγματικό όμω ζήτημα, και εκεί πάντα λέμε ότι θέλουμε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη-μέλη, είναι το ζήτημα τη ορθή εφαρμογή, υλοποίηση. Δεν είναι η μεταφορά. Γιατί εκεί μπορεί κάποιε διαδικασίε να καθυστερούν κάπω, αλλά συγκριτικά είναι πολύ λιγότερο σημαντικό ζήτημα από ότι αυτό τη ορθή υλοποίηση τη οδηγία. Είχατε κάτι επιπλέον. όταν είναι να στείλουμε τις επίσημες επιστολές Μπορώ να σα δώσω τις μερμήνες που ποτέ στείλαμε τι επίσημες επιστολέ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο ενδιαφέρον για σας, Είναι πολύ λεπτομέρεια. Η πρόεδρος Δεν ξέρω αν θέλει να επανέλθει κανείς. Οι ερωτήσεις που άκουσα εγώ από τα μέλη μου δίνουν την εντύπωση πω θα ήθελαν περισσότερο σαφή εικόνα για το ποιες είναι αυτές οι δημόσιες αρχές οι οποίες αντιμετωπίζουν συχνά διαμαρτυρίες και προβλήματα. Είπατε ότι μπορεί να μην είναι σωστή λύση αυτή ενός ε, πίνακα των ε, κακών επιδόσεων μιας μαύρης λίστας, αλλά θα ήταν καλό να βοηθήσουμε και τους συναδέλφους να καταλάβουν περισσότερο ποια είναι η κατάσταση και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε μια διαδικασία, δεν θα πω καταγγελίας, αλλά εν πάση περιπτώσει να ρίχνουμε φως στις καταστάσεις και να βλέπουμε ποια είναι τα κράτη αυτά που τακτικά παραβαίνουν τους όρους της οδηγίας και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και την ενημέρωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που λένε οι συνάδελφοι εδώ είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση σε επίπεδο κρατών μελών ή τοπικό επίπεδο. Μπορεί να μας λέτε ότι κάνει διαφορά η Επιτροπή, αλλά ίσως θα πρέπει να σας απασχολήσει εσωτερικά το θέμα της βελτίωσης. Και πάλι για να μιλήσω για τις ε, παραβάσεις. Ένας τρόπος να το αντιμετωπίσετε είναι, όπως είπε ο κύριος Φαπ, να ενθαρρυνθούν οι αρχές να μην προβούν σε παράβαση, να μην ξεκινήσει η παράβαση. Και άρα θα ήταν καλό να είναι γνωστό ποιο κράτος ή τι είδου κράτος ή με ποιού όρους, σε ποιον τομέα, τακτικά φερειπήρ στον χώρο της δημόσιας υγείας, των μεταφορών, που διαπιστώνεται τις ε, καθυστερήσεις, τις πληρωμές. So I would suggest the may want to follow up with you Θέλετε να ξαναπάρει το λόγο. Ε, ναι, ε, κλείνοντας να πω τα εξής. Το είπα και πριν, οι βασικές χώρες στις οποίες υπάρχουν προβλήματα σε όλους τους τομείς. Ο τομέας υγείας προφανώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ε, είναι η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό. Έχουμε πολλές αποδείξεις για το ότι δεν λειτουργεί η εφαρμογή της οδηγίας. Υπάρχει μια ε, κυβερνητική οργάνωση ε, η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή και το μέσο όρο καθυστέρησης και τα απορίσματά της είναι παρόμοια με τα δικά μας. Ε, τώρα, αν έχετε όμως κάποια πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, κάποια πιο, συγκε, κάποιες πιο συγκεκριμένες καταγγελίες ή θέματα, ε, να σας ενημερώσουμε διμερώς ο Κώστας Ανδρόπουλος ε, εξακολουθεί να είναι μαζί μας ότι αν και οπότε αν θέλετε να σας απαντήσει κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο μιλήστε μαζί του. Okay, so I'm going to ask the to make... Θα ήθελα να ζητήσω από τη γραμματεία να έρθει σε επαφή με τα μέλη τα οποία έλαβαν το λόγο σήμερα για να ε, δούμε ποια λεπτομερή, ποιες λεπτομερείς ε, πληροφορίες χρειάζονται και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας προκειμένου να πάρουμε αυτές τις πολύ συγκεκριμένες ε, πληροφορίες, ανακλάδο κλπ. Είναι προφανές ότι πολλά μέλη ε, ενδιαφέρονται να δουν τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε περαιτέρω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. getting me confusing. Right, let's. Um, Right, so the first um, uh, vote this morning is... Η πρώτη ψηφοφορία σήμερα το πρωί αφορά την έκθεση για τα όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά οχήματα. δεν έχει να πει κάτι ο εισηγητή, να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. οποίο ε, είναι υπέρ, πώ είναι κατά. Δεν έχει κατάλογο ψηφοφορίας η Πρόεδρος. Ο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μαζί από 36 μέχρι 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ με προφορική τροπολογία τι έχετε μπροστά σας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 λέγεται ψηφοφορία συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ απο, κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μαζική ψηφοφορία 10, 11, 12 και προφορική 13 και 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 και 53 αποσύρονται 54 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά να το ελέγξουμε εγκρίνεται 16 τίποτα, 17-18 εγκρίνεται, 55 αποσύρεται, 19 με προφορική τρόπο λέγει υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 21 και 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 20 δεν ψηφίζεται, 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 23 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 24 δεν γίνεται ψηφοφόρια. 57 ε, ε, εγκρίνεται. 57. Περνάμε σε επιλογές σκέψεις. 1. Υπερκατάποχες εγκρίνεται. 2. Υπερκατάποχες εγκρίνεται. εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές Ελεγ... αναελέγξουμε ηλεκτρονικά ακόμα δύο ψήφοι απορρίπτεται 37 ε, υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 28 να ελέγξουμε την 27 νομίζω ότι είναι η ίδια πλειοψηφία η κάρτα που βρίσκεται εδώ αλλά δεν αναγνωρίζεται από κανένα από τα μηχανήματα 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 απορρίπτεται 32 απορρίπτεται 33 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και για την όλη έκθεση για την τελική έκθεση με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 30 υπέρ, 2 κατά και 4 αποχές. Πολλά συγχαρητήρια γύρι. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Το επόμενο ψηφοφορία είναι η έκθεση του Νικολαντάτη για την πιθανή επέκταση της προστασίας γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Ντάντη, θα θέλατε να πείτε κάτι για να ξεκινήσουμε. Okay, amendment one. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ κατά εγκρίνεται, συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 11 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ Πρόκειται για διαγραφή εδώ. Άρα δεν είναι κομμάτι της συμβαστικής υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται συμβαστική Β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική δ δέλτα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 32 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται 33 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται H συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ όχι ζητώ συγγνώμη λέει ο πρόεδρος έχουν καταπέσει οι 62 και 63 δηλαδή συμβαστική Άι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται J συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές 70 λέει η πρόεδρος 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 αποσύρθηκε 82 προκτήρια διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται L συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 88 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για το σύνολο της νομοδότησης παρακαλώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγκρίνεται λοιπόν 32 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά, αποχή 1. Και συγχαρητήρια Νίκολα. Έχουμε λίγο καθυστερήσει. Έχουμε ένα μικρό περιθώριο χρόνου λοιπόν ε, και μια και είχαμε πει ότι θα σας ενημέρωνα για τον τριμερή διάλογο ε, μια και δεν ήμουν χτες εδώ, μπορώ να σας πω τα εξής. Έχουμε αρμοδιότητα Επιτροπής για τα, ε, για το, για τα προϊόντα, για την τελική χρήση των προϊόντων και είχα αναλάβει ως διάδοχο του Malcolm Harbour τη θέση του στον τριμερή διαλογό. Ήταν πολύ σκληρέ οι διαπραγματεύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και οι εισηγητέ για τη βοήθεια και τις καλές ιδέες που προσέφεραν ώστε να προχωρήσουμε. Στον πρώτο τριμερή διάλογο η Προεδρία μας διαβεβαίωσε ότι θα μας κάνει μια σαφή πρόταση για τα προϊόντα του χρήστη ενσωματώνοντας τα ε, κεφάλαια για τα τέλη. Δια, ε, περιαγωγής χωρίς να περιμένει την τελική εκδοχή του USD. Τις τελευταίες μόνο εβδομάδες σημειώθηκε πρόοδος όμως στον τριμερή διάλογο για τα δικαιώματα του τελικού χρήστη. Για την περιαγωγή η Προεδρία δέχθηκε τις περισσότερες από τις προτάσεις και απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα κύριο ζήτημα δηλαδή ιδιαίτερα πριν να κλείσει το θέμα του Ρώμη, πριν να λήξει δηλαδή το τέλος περιαγωγής, να ενημερώνεται ο χρήστης για ένα για το μέγεθος του πακέτου που του και όταν πρόκειται να περάσει ε, σε ένα πιο ακριβό επίπεδο τιμών να του έρχεται ένα μήνυμα. Διαφάνεια, διαφάνεια λοιπόν. Οι διατάξει διαφάνειας γίνονται διεδεκτές. Αλλά εμείς διεκδικούμε και έλεγχο κατανάλωσης κυρίως ε, με ενημέρωση το, μέσω ε, SMS του καταναλωτή για το τιμολόγιο στο οποίο έχει περάσει. Για τα δικαιώματα του τελικού χρήστη αντιστέκεται περισσότερο το Συμβούλιο. Θα γίνει άλλη μια συνεδρίαση των σκιωδών και τριμερής διάλογος την επόμενη εβδομάδα. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η δυνατότητα ο τελικός κρίστης να, να ακυρώνει, να τροποποιεί το, τη σύμβασή του εάν δεν του προσφέρονται οι υπηρεσίες στην ταχύτητα με την οποία είχαν προβληθεί διαφημιστικά. Άρα για, το, για τα δικαιώματα τελικού χρήστη στην περιαγωγή είμαστε ικανοποιημένοι, όμως για την χρήση του ίντερνετ ε, όχι τόσο. Άλλη μια συνεδρίαση λοιπόν σκιωδών συγκητών. Θα συζητήσουμε μαζί λύσεις για να καλύψουμε το χάσμα μεταξύ των θεσιών ημών και εκείνων, ώστε να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον μεγαλύτερη διαφάνεια για το χρήστη, να γνωρίζει τι του προσφέρεται και τι μπορεί να κάνει εάν δεν είναι η υπηρεσία στο ύψος που του είχαν υποσχεθεί, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ατελείωτες ήταν οι ώρες των διαπραγματεύσεων η γραμματεία, οφείλω να πω, η γραμματεία της Επιτροπής μας ε, μας προσέφερε τεράστια βοήθεια και πολύ αποτελεσματική. Σας ευχαριστούμε. Έχετε ερωτήσεις για αυτό το θέμα? On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 is you just vote too fast. So I'm going to suggest we... Ε, ψηφίσαμε υπερβολικά γρήγορα. Ε, τελειώσαμε τι ψηφοφορίες πολύ πιο νωρίς από ό,τι περιμέναμε. Ε, είμαστε πάρα πολύ καλά οργανωμένοι, <laughs> αλλά δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την ε, διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων μέχρι ότου έρθουν οι εμπειρογνώμονε. Γιατί αυτοί θα μας παρουσιάσουν τα ενημερωτικά σημειώματα. Οπότε, προτείνω να διακόψουμε 15 λεπτά και να ελπίζω, και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να ξεκινήσουμε στις 10 και 20, δηλαδή πριν από τις 10.30 που ήταν ο προγραμματισμένος χρόνος έναρξης. Μας ενημερώνουν ότι θα είναι εδώ σε 10 λεπτά, οπότε θα ξεκινήσουμε στις 10 και 4. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Περνάμε στην ε, TTIP, τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων. Ε, έχουμε σημειώματα, τρία εμνημερωτικά σημειώματα. Ε, η συγγραφή συγγραφείς είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Στίβεν Βίλκοκ, επικεφαλής του LSE στην Μονάδα Διεθνούς Εμπορίου, Προστασία καταναλωτών, η κυρία Μπάρμπαρα Χόλσον, ε, επίσης από το LSE, ερευνήτρια, και ο Πομακρόν φίλος της Επιτροπής μας, ε, ο οποίος θα μας ε, παρουσιάσει το θέμα των προτύπων. Οι βασικοί διαπραγματευτέ τη Κομισιόν έχουν προσκληθεί να απαντήσουν σε ερωτήσει, θα έρθουν αργότερα. κύριος Γουλκοκ, ε, η, ο, η, ομάδα του κ. Γουλκοκ θα φτάσει λίγο καθυστερημένη και θα απαντήσει ερωτήσει αν δεν μπορούν να απαντήσουν οι παρόντες. Ο κ. Κόσμος είναι επίσης μαζί μας εδώ, που επίσης έχει εργαστεί για τα ενημερωτικά σημειώματα. Ε, δέκα λεπτά κάθε παρουσίαση παρακαλώ. Τρεις παρουσιάσεις και μετά ερωτήσεις ε, από τους παρόντες αν είναι δυνατόν. Παρακαλώ πολύ 10 λεπτά η κάθε παρουσίαση, ο λόγος στον κύριο Γουλκοκ. Um, Θα παρουσιάσω τις δημόσιες προμήθειες. Εγώ. Πρώτα μια καταρχάς από, το... από τη μελέτη μας. Οι δημόσιες προμήθειες ε, είναι ένα ζήτημα της TTIP όπου έχει επιθετικό όπως λέμε συμφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή αποσκοπεί στο να επιτύχει περισσότερα κυρίως όσον αφορά την κάλυψη των προμηθειών σε κρατικό επίπεδο και επίπεδο πολιτιών, ε, πόλεων μάλλον στις ε, πολιτιών και πόλεων στις ΗΠΑ. Πρόκειται και μια λειτουργική αρμοδιότητα, δηλαδή πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο οι de όσο και οι de facto φραγμοί στον ανταγωνισμό. Αυτό σημαίνει ρητά νομοθετημένες προτιμήσεις υπέρ των ε, εγχωρίων προμηθευτών, αλλά και άλλες οι οποίες προκύπτουν μόνο από την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας και όχι από τους κανόνες. Αυτό μπορούμε να το έχουμε υπόψη και πρέπει να το έχουμε υπόψη νομικές de jure δηλαδή, αλλά και de facto πτυχές. Ένα άλλο σημείο σημαντικό στις διαπραγματεύσει έχει να κάνει με την βελτίωση της ε, ουσιαστικής διαφάνειας. Το να γνωρίζουμε δηλαδή τι συμβαίνει, τι ισχύει στις ε, προμήθειες. Ποιες είναι οι διαδικασίες τους, πότε δημοσιεύονται οι προσκλήσεις και εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Όλα αυτά τα ζητήματα θα τα αναπτύξω στη συνέχεια. Μας ζητήθηκε λοιπόν να εξηγήσουμε πώς μπορεί να επηρεάζονται οι γενικές διατάξεις περί εμπορίου σε επίπεδο ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορεί η TTIP να αλλάξει κάτι. Γιατί ξέρετε ότι και η συμφωνία με τον Καναδά, η ΣΥΤΑ, είχε συμπεριλάβει το ζήτημα των δημοσίων προμηθειών. Ήταν άλλωστε κύριο στοιχείο οι δημόσιες προμήθειες στην ΣΥΤΑ και η κάλυψη επίσης των ε, ε, προμηθειών σε επίπεδο επαρχίας και τοπικών αρχών. Αυτό το επέτυχε η ΣΥΤΑ. Άρα έχουμε ένα πολύ καλό προηγούμενο σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις TIP. Θα αναφερθώ επίσης στις προκλήσεις και μια από τις κύριες προκλήσεις είναι στην όλη αυτή τη συζήτηση να πείσουμε τα τοπικά κοινοβούλια των ΗΠΑ να ανοίξουν τις ε, προμήθειές τους στις ξένες αγορές. Εδώ είναι ένα ζήτημα ε, δομής πολιτιακής, γιατί το USGL, ξέρετε, οι διαπραγματευτές εκ μέρους των ΗΠΑ δεν μπορούν να δεσμευτούν δεδομένου ότι αυτό το ζήτημα των δημοσίων προμηθειών ανήκει στις αρμοδιότητες των πολιτιών και όχι του Ομοσπονδιακού κράτους. Το 13% του ΑΕΠ λοιπόν στην αγορά των ΗΠΑ καλύπτεται από τις ε, προμήθειες. 65% σε υπό ομοσπονδιακό επίπεδο, δηλαδή στα ομοσπονδα κρατήδια. Και στην πραγματικότητα έχουμε πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Αυτά τα ποσά δηλαδή που βλέπετε δεν είναι ακριβή, είναι υπερβολικά. 4% ουσιαστικά του ΑΕΠ. Αλλά πάλι είναι σημαντικό μερίδιο για οποιαδήποτε αγορά. ωφελούνται κυρίως εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα, εάν προκύψουν ε, κατά τρόπο επιτυχή διαπραγματεύσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση έμεσα στις αγορές, έμεσα όπως λέμε, στον κλάδο μας, δηλαδή με τις επενδύσεις τοπική οικονομία και την ε, προμήθεια στις ε, δημόσιες υπηρεσίες και αρχές μέσω αυτών των τους, ενώ μια μικρομεσαία επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να επενδύσει στην τοπική αγορά. Άλλοι τομείς που μπορεί να ωφεληθούν, οι μεταφορές, παραδείγματι, όπου δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι αγορές, σιδηροδρομικά, λεωφορεία και το καθεξής. Ο κατασκευαστικός κλάδος, και μάλιστα είναι και οι δύο κλάδοι, και των μεταφορών και των κατασκευών, κλάδες ο οποίος έχει ιδιαίτερη ευρωστία η ευρωπαϊκή οικονομία. Οφελείται δε και ο φορολογούμενος γιατί αξιοποιούνται καλύτερα οι δημόσιοι πόροι. Με περισσότερη διαφάνεια έχουμε περισσότερη ακαιρεότητα όπως λέμε στις δημόσιες προμήθειες, δηλαδή περιορίζεται ε, το περιθώριο για καταχρήσεις στις δημόσιες συμβάσεις και θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στη φύση των φραγμών. Οι υφιστάμενοι φραγμοί λοιπόν είναι οι de jure, οι υφιστάμενες νομικές προτιμήσεις. Αυτό που λέμε buy America ή buy American, αγοράζει τα αμερικανικά προϊόντα. Όταν υπάρχουν ρητές προτιμήσεις για παραγωγού Αμερικανού σε ορισμένε περιπτώσει. Αν θέλετε θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειε στη συνέχεια στι ερωταπαντήσει. Επίσης, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν σε μειονότητε. Σημαντικές λοιπόν εξαιρέσεις και εμπόδια αλλά επίσης πολύ σημαντικές είναι και οι de facto προτιμήσεις που θα εκθέσω στο κεφάλαιο για τη διαφάνεια. Η διαπραγμάτευση αφορά την κάλυψη ορισμένων τομέων σαν να ήταν εθνικός ο προμηθευτής, δηλαδή να μην υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση όταν καλύπτονται ορισμένες προδιαγραφές για τις ε, κρατικές αρχές, πολιτιακές αρχές και επαρχιακές αρχές. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε έναν προτιμησιακό καθεστώς για τις δημόσιες προμήθειες που καλύπτει κάθε επίπεδο διακυβέρνησης, κεντρική, περιφερειακή, τοπική, ε, δημόσιες υπηρεσίες. Ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ένα ομοσπονδιακό επίπεδο κανόνων ε, για τις δημόσιες προμήθειες που αφορά μόνο το Ομοσπονδιακό κράτος και τις προμήθειες που μπορεί να αφορούν λίγες πολιτείες όταν αυτές καλύπτονται από τις σχετικές συμφωνίες δημοσίων προμηθειών. Ενώ άλλες δημόσιες προμήθειες των πολιτιών ή των πόλεων δεν ακολουθούν ένα ενιαίο σύστημα δημοσίων προμηθειών. Άρα οι διαδικασίε μέσα από τι οποίε πρέπει να περάσει ο προμηθευτή ποικίλουν από τη μία πολιτεία στην άλλη και από τη μία πόλη ακόμη στην άλλη. Εδώ λοιπόν τίθεται το ζήτημα τη διαφάνεια, γιατί πάλι μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση τη Ευρώπη, αν προσπαθεί να έχει πρόσβαση στην Αμερικανική αγορά, θα πρέπει και να γνωρίζει πώ ε, λειτουργούν οι διαδικασίε στην Καλιφόρνια, συγκεκριμένα το Λο Άντζελε, αλλά πρέπει να έχει υπόψη και τις διαδικασίες που ισχύουν στο Χιούστον του Τέξα για τι δημόσιε προμηθείε και αυτέ μπορεί να διαφέρουν πολύ. Άρα, η απέτηση της διαφάνειας, η προϋπόθεση της κοινοποίηση των διαδικασιών, της δημοσιοποίησης των διαδικασιών και των όρων είναι πάρα πολύ σημαντική ε, προϋπόθεση για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι φραγμοί. Και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η κάλυψη των καθεστώτων δημοσίων προμηθειών στηρίζεται σε αμοιβαία διαπραγμάτευση. Και αυτό ισχύει και ότι υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο ΠΟΕ για τις δημόσιες προμήθειες. Στηρίζονται στις διμερείς αμοιβές διαπραγματεύσεις στις δημόσιες προμήθειες. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχουν διαπραγματευτεί επί δεκαετίες την αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές των δημοσίων προμηθειών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε όμως δεν καλύπτουν το, ε, τις προμήθειες, δημόσιες προμήθειες σε επίπεδο πολιτιών ή σε επίπεδο πόλεων. Και αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρακρατήσει την κάλυψη ε, ορισμένου επίπεδου δημοσίων προμηθειών εντό Ευρωπαϊκή Ένωση για προμηθευτέ από τι ΗΠΑ. Διαφάνεια. Τελευταία μου παρατήρηση. Η διαφάνεια είναι εν πολλής εξίσου σημαντική με την καταπολέμηση των de facto φραγμών. Προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σημαντικό βαθμό διαφάνεια γιατί έχει ένα ομοιόμορφο καθεστώς με διαδικασίες ε, ίδιες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξαρτήτως του επίπεδου των προμηθειών. Αυτό όμως δεν ισχύει ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και αυτό καθιστά λιγότερο διαφανή την αγορά των Ηνωμένων Πολιτείων. Προκλήσεις. Που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στις διαπραγματεύσεις. Πρώτα απ' όλα ότι δεν έχει η διαπραγματευτική ομάδα την αρμοδιότητα για να καλύψει πολιτείες και λοιπούς, ε, λοιπές κρατικές οντότητες για να προσαρμοστούν στο επίπεδο αυτών των διαπραγματεύσεων, στις απαιτήσεις των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να τις πείσει λοιπόν και επίσης τα νομοθετικά όργανα στις πολιτείες δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένα να ε, δώσουν ε, χρήμα του Αμερικανού φορολογουμένου για να χρηματοδοτήσουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, σε απλά λόγια οικονομικών όρων. Άρα είναι δύσκολο να ανοίξουν αυτές οι αγορές για τις δημόσιες προμήθειες σε επίπεδο πολιτείας και πόλεως. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι Υπήρξαν μέχρι πρόσφατα ε, διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τις Δημόσιες προμήθειες, του ΠΟΕ. Και εκεί έχει γίνει ένα μεγάλο μερίδιο της δουλειάς. Και σημαντικό μερίδιο. Και άρα ναι, μπορεί να έχει σοβαρό και επιθετικό, όπως λέμε, συμφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι προκλήσεις για τους Αμερικανούς είναι επίσης σημαντικές. Πρέπει να ανοίξουν αγορές τους. Προοπτικές. Οι προοπτικές θα εξαρτηθούν ε, από την πρόοδο της δέσμης μέτρων. Δηλαδή, πρόοδο στις δημόσιες προμήθειες δεν αναμένεται να δούμε εάν δεν υπάρχει αντίστοιχα πρόοδο σε άλλους τομείς της TTIP. Και αναμένεται διασύνδεση, όπως συμβαίνει πολύ συχνά μεταξύ διαφόρων θεμάτων. Κατά πόσο πιθανότητα θα γίνει μάλιστα, θα καταστεί μάλιστα κομμάτι ε, το θέμα των δημοσίων προμηθειών μια ζώσα συμφωνία με την έννοια ότι το τελικό κείμενο θα αποτελέσει μόνο ε, ένα βήμα στην διαδικασία ανοίγματο των δημοσίων προμηθειών που θα πρέπει να συνεχιστεί μετά. Η βελτίωση των ε, βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τι δημόσιες προμήθειες άλλωστε και ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, πολιτιακέ αρχές θα περάσει μέσα από το να πισθούν αυτές ότι είναι προς το συμφέρον τους να προχωρήσουν σαν να είχε κλείσει μια ολόκληρη συμφωνία. Και θα σταματήσω εδώ, Πρόεδρε. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να ακούσετε όλες τις, πα, τις παρουσιάσεις αμέσως. Η Πρόεδρος, κοιτάω τους αδέλφους, θέλετε να ακούσετε και τις τρεις παρουσιάσεις και μετά να κάνουμε τις ερωταποντήσεις. Ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά θα ακούσουμε και τους άλλους ομιλητές. Η Βάρβαρα έχει πολύ ενδιαφέρον βιογραφικό, έχει εργαστεί και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. So, good morning, ladies and gentlemen. My name is Petros Kuzmu. Ονομάζομαι Πέτρος Κούσμου. Είμαι από τον Καναδά, αν δεν καταλάβατε την προφορά μου. Η Μπάρμπαρα ε, είμαστε από το, και εγώ είμαστε από το LSE ε, για το Τμήμα Προστασίας Καταναλωτή. Θα συζητήσουμε το θέμα, ε, του, το θέμα αυτό προστασίας καταναλωτή σε σχέση με την TTIP. Τρεις τριπλός ο στόχος μας. Πρώτον, να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε σε εθνιστικό επίπεδο ε, δεύτερον, να δούμε τι συνεπάγεται τι για, την για την προστασία του καταναλωτή ε, και τρίτον, τι συνεπάγεται ε, σε ό,τι αφορά την, τις εξουσίες του Κοινοβουλίου. Τα βασικά μας πορίσματα είναι ότι οι εξουσίες του Κοινοβουλίου δεν πρόκειται να επηρεαστούν από την TTIP. Παρ' όλα αυτά, προτείνουμε το Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι οι, προ, οι προτεραιότητες θα ληφθούν υπόψη στην συνεργασία. Ε, έχουμε διαφορετικές ε, θεσμικές διαδικασίες και διαφορετικές φιλοσοφίες και αυτό είναι στις δύο μεριές του Ατλαντικού και αυτό είναι, δημιουργεί ε, κάποια προβλήματα. Ε, εκτίμηση, τελική εκτίμηση όμως του αντικτύπου θα μπορεί να γίνει μόνο αφού ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ε, γιατί η συνεργασία σε ρυθμιστικά θέματα είναι τόσο σημαντική στην TTIP. Πρώτον, τα περισσότερα ωφέλη από την TTIP θα προκύψουν χάρη στην ε, βελτίωση της συνεργασίας και όχι τόσο πολύ εξαιτίας της μείωσης των δασμών δασμοί που βρίσκονται σε επίπεδο 45% ε, και τα ωφέλη που θα προκύψουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός της μείωσης των δασμών θα είναι 70-120 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Στη, σε ό,τι αφορά μείωση των δασμών, ως τώρα υπήρχε Συγγνώμη, ε, η βελτίωση τη συνεργασία σε εθνιστικό επίπεδο ήταν δύσκολη στο παρελθόν εξαιτία του ότι έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα. Δεύτερον, γιατί δεν έχουμε αρκετή πολιτική στήριξη στη διαδικασία αυτή, στο, δεν είχαμε στο παρελθόν. Και τρίτον, πολύ συχνά οι νομοθέτε φοβούνται θα χάσουν εξουσία. Ε, στην οικονομική συνασία του οικονομική συνασία του 1998 ε, ε, έγιναν προσπάθειες για να περάσει μια αναγνώριση αλλά προέκυψαν πολλά εμπόδια. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς ομιλήτρια. Ε, ποιες ε, είναι οι επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τρεις ε, δυνατότητες για την συνεργασία αυτή. Πρώτον, να διευρυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις ρυθμιστικές αρχές των δύο περιοχών. Δεύτερον, αμοιβαία αναγνώριση ή ισοτιμία. Είναι περίπου το ίδιο πράγμα, αλλά είναι διαφορετικό ο τρόπος κάθε μιας από τις δύο αυτές δυνατότητες. Και η τρίτη πρόταση είναι η εναρμόνιση ή απλοποίηση. Το θέμα όμως θα είναι αν η εναρμόνιση θα γίνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Ε, παρόλο ότι υπάρχουν φόβοι ότι θα κινηθούμε προς τα κάτω με την εναρμόνιση, υπάρχουν δυνατότητες να κινηθούμε και προς τα πάνω. With regards to how regulatory cooperation will... Ε, το πώς θα λάβει η χώρα η ρυθμιστική ε, συνεργασία. Ε, η, να έχουμε στο μυαλά μας ότι θα είναι μια ζώστα συμφωνία. Όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, εκεί θα ξεκινήσει η διαδικασία της ρυθμιστικής συνεργασίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ο στόχος των διαπραγματευτών είναι να δημιουργηθούν, να θεσπιστούν διαδικασίες έτσι ώστε οι συνεργασία να γίνει σωστά. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να είναι διαφανές ε, αλλά και αποτελεσματικό. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν προτείνει τη δημιουργία ενός σώματος, ενός φορέα συνεργασίας, ε, ρυθμιστικής συνεργασίας ε, ο οποίος θα συντονίζει την συνεργασία σε διάφορους τομείς σε ρυθμιστικό επίπεδο θα είναι ε, το βασικός φορέας ε, ο οποίος θα ρυθμίζει αυτή τη συνεργασία αν εγκριθεί η πρόταση της Κομισιόν. Ε, στόχος μας ήταν να αξιολογήσουμε το πώς θα επηρεαστεί η προστασία του κατανοητή και η εξουσία του κοινοβουλίου σε αριθμιστικά θέματα. Ε, μειωμένα κόστη ε, και πιο ανταγωνιστικές αγορές ε, είναι ένα από τα, τις, μία από τις, τα βασικά ωφέλη. Η, θα μειωθούν οι έλεγχοι στα σύνορα, θα αυξηθεί η, το εμπόριο και η πρόσβαση αγορές. Δεύτερον, από κοινού θα μπορέσουμε να τροποποιήσουμε και να διαμορφώσουμε τους διεθνείς κανόνες εμπορίου και πρότυπων και τα διεθνή πρότυπα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ε, σύγκληση, κάτι βέβαια, που θα βοηθούσε για το εμπορικό σύστημα. Τρίτον, τρίτη ευκαιρία, τρίτο όφελος, αύξηση του ανταγωνισμού, μείωση των τιμών και βελτίωση της ποικιλία που προσφέρεται στους καταναλωτές σε ό,τι αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Επιπλέον, η αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών θα βελτιώσει τις, πολιτικέ τις πολιτικές υπέρ του καταναλωτή. Μάλιστα μπορεί οι ρυθμίσει TTIP να γενικευτούν στο παγκόσμιο εμπόριο και αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο. Βέβαια, η αύξηση του ανταγωνισμού των αγορών δεν σημαίνει ε, ελάχιστο κοινό θα πρέπει να δούμε πού χρειάζονται παρεμβάσεις και πού ο συντονισμός μπορεί να οδηγήσει σε ωφέλη. Επίσης υπάρχει η ευκαιρία αυτές οι διαπραγματεύσεις να δώσουν εξωτερική όθηση στην αλλαγή των εσωτερικών πολιτικών. Βέβαια με τις μεγάλες, προκλήσεις, με τις μεγάλες υποσχέσεις έρχονται και μεγάλες προκλήσεις. Στην μελέτη μας υπογραμμίζουμε τέσσερις προκλήσεις βασικά. σε ό,τι αφορά την προστασία του καταναλωτή. Πρώτον, είναι δύσκολο να συμφιλειώσουμε τι δύο διαφορετικέ ρυθμιστικέ φιλοσοφίε ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί ε, την ε, αρχή τη προφύλαξη, οι ΗΠΑ ε, ακολουθούν μια πιο επιστημονική προσέγγιση. Οπότε η ρυθμιστική συνεργασία σε ορισμένου τομεί θα είναι πιο δύσκολη, πιο επιφανειακή. Ε, η ανταλλαγή πληροφοριών, για παράδειγμα, μπορεί να είναι πιο εύκολη στον τομέα των χημικών, τη χημική βιομηχανία. Δεύτερον, θα πρέπει να βρούμε πού θα λειτουργήσει καλύτερα η συνεργασία ε, και ποιε θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητέ μα. Αφού αυτή η συμφωνία, η συνεργασία ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα γίνουν οι κατάλληλε επιλογέ στους κατάλληλους τομείς έτσι ώστε εκεί που πιο πολύ χρειάζεται και μπορεί να λειτουργήσει να εφαρμοστεί η συνεργασία. Τρίτον, ε, η διαδικασία θα πρέπει να είναι η πιο κατάλληλη. Θα πρέπει το πλαίσιο της συνεργασία να διασφαλίζει ότι θα γίνονται συνεχείς προσπάθειες και ότι ο, ο φορέας ο οποίος προτείνουμε να δημιουργηθεί ε, θα λειτουργεί σωστά και θα η, το, η εργασία του θα αντανακλά τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτον, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι εξουσίες του Κοινοβουλίου θα προστατευτούν. Από ό,τι φαίνεται όμως ως τώρα, από το κείμενο της Κομισιόν φαίνεται ότι προστατεύονται. Το όργανο ε, ρυθμιστικής συνεργασίας δεν θα έχει εξουσίες οι οποίες να περιορίζουν τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή θα έχει τον τελευταίο λόγο. Λοιπόν, στη μελέτη μας ε, κάναμε μελέτες περιπτώσεων σε τέσσερις τομείς που θα παρουσιάσουμε συντομία. Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας θα υποφεληθεί από τη ρυθμιστική σύγκληση, ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για το μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο κίνητρο αντιμετωπίζοντα τα αριθμιστικά κόστη για διάφορα προϊόντα, τι μεθόδου ε, δοκιμών. Ε, θα υπάρχουν διαφορετικοί κανονισμοί, αλλά διασφαλίζουν παρόμοιο επίπεδο ασφάλειας. Αλλά για πολλούς κανονισμούς ε, υπάρχει δυνατότητα αμοιβέ αναγνώριση. Αυτό συνάδει με την πρότασή τη ε, Επιτροπής ε, το Μάιο του 2014 που διατυπώνει ένα τετραπλό στόχο ανάπτυξη μιας μεθοδολογικής προσέγγισης και, και κριτηρίων για την αναγνώριση της αντιστοιχίας και κάποια συνεργασία που θα οδηγήσει στην υιοθέτηση κοινών προτύπων. One of the other case studies. Μια από τις άλλες μελέτες περιπτώσεις όπου τάσαμε ήταν ο τομέας ε, των τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών και θεωρήσαμε ότι υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας ε, στον τομέα της πληροφορικής αλλά κάποιοι τομείς είναι ενισχυτικοί όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Οι καταναλωτές ε, θα υποφεληθούν από την αυξημένη ρυθμιστική συνεργασία σε διάφορα τομείς όπως η ηλεκτρονική επισήμανση και άλλοι. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει ως αποτέλεσμα να μειώσουν το δαπάνες τους και να... αυτό θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές. Ένα πρόβλημα είναι η ελεύθερη ροή δεδομένων και η Ευρώπη δεν θέλει να διαπραγματευτεί το απόρριτο των δεδομένων. Η δεν θέλουν να αλλάξουν ιδιαίτερα τα μέτρα τους. Θέλουν να υπάρξουν κάποια μέτρα σε ένα κεφάλαιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά υφίστανται πίεση από διάφορους παράγοντες στη ΣΥΠΑ. Η ΣΥΤΑ αποτελεί καλό μοντέλο για τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές όσον αφορά τα μέτρα Προστασία των δεδομένων και απλά ζητείτε να σέβονται και τα δύο μέρη τα σημερινά πρότυπα που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο. Ε, Για να κλείσουμε. Όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, προτείνουμε η ρυθμιστική κυριαρχία ξέρετε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα επηρεαστεί από την TTIP. Θα είναι μια ζώσα συμφωνία, δηλαδή ένας διμερής μηχανισμός συνεργασίας. Συμμορφώνται με τους σημερινού μηχανισμούς ε, δημοκρατικού και πολιτικού ελέγχου. Εφόσον υιοθετηθεί η πρόταση της Κομισιόν, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να είναι ο εξή. Θα ασχολείται με οποιαδήποτε δράση που απαιτεί νομοθετική αλλαγή, θα διασφαλίζει ότι το όργανο ρυθμιστικής συνεργασίας θα είναι διαφανές και θα εξετάζει τις ε, προτεραιότητες ε, του ετήσιου προγράμματος ρυθμιστικής ε, συνεργασίας ώστε να διασφαλίζει ότι αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες και το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Εγώ διάβασα ολόκληρο ε, την έκδοση καθώς και την παρουσίασή σας. Ε, όλα τα έγγραφα αυτά υπάρχουν διαθέσιμα επίσης και ηλεκτρονικά. Και ε, θα τα κοινοποιήσουμε βεβαίω μεγάλη ευχαριστήση με τι χιλιάδε άτομα που επικοινώνησαν μαζί μα για τα ζητήματα αυτά. Επόμενο ομιλητή ο Ζακ Πέλκμαν που θα μα παρουσιάσει την έκθεση του για τα πρότυπα. Ευχαριστούμε Ζακ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, αξιότιμα μέλη, με μεγάλη μου χαρά θα σας παρουσιάσω την πυρήνα του TTIP. Θα μιλήσουμε επιτέλους ε, για τα πράγματα ως έχουν. Θα σας δώσω κάποια συμπεράσματα και μετά θα μπω στην ουσία, διότι δεν μιλάμε απλά για τα ε, τεχνικούς φραγμούς του εμπόριο και τα πρότυπα. Μιλάμε για κάτι πολυτεχνικό, όχι από άψη μηχανικής. Το πρώτο που θέλω να πω είναι, όπως είπα, μιλάμε για το ε, ε, νουσία του TTIP. Δεύτερον, δεν θα συμβούν και πολλά αν οι ΙΠΑ χρησιμοποιήσουν ε, το template που έλεγαν ότι θα χρησιμοποιούσαν. υπάρχει ένα κεφάλαιο TBT και είναι αδύναμο. Συμφωνώ με την Κορέα. Ε, το τρίτο είναι το TBT ε, εντός του TTIP δημιουργεί πέντε συστημικά ερωτήματα που θα αναφέρω ε, ε, σύντομα. Πρώτα, τα συστήματα τυποποίησης είναι διαφορετικά. Δεύτερον, όχι επαρκής χρήση των προτύπων το ISO και IC στην Αμερική. Τρίτον, ο, τρίπος που σχετι... ο τρόπος που σχετίζονται τα πρότυπα με τους κανονισμούς. Συχνά συγχαίουμε αυτούς τους όρους. Ε, ένα πρότυπο για αυτοκίνητα δεν είναι πρότυπο, είναι ε, κανονισμός, είναι ρύθμιση. Τέσσερα, η αξιολόγηση συμμόρφωσης και πέντε, το κατά πόσο θα επιτρέπεται ή όχι θα επιτρέπεται ή όχι ανταγωνιστικά πρότυπα στις ε, κατάρθαν αγορές. Ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο ε, χαλαρή η κατάσταση. Μπορείς να προχωρήσεις παρακαλώ της Όχι, όχι, γιατί ακόμα δεν έχω μπει στο θέμα της διαφάνειας. Λοιπόν, τι είναι η TTIP, τι βλέπετε εδώ για όποιον ενδιαφέρεται η ουσία της βλέπετε στο μέσον το ρυθμιστικό της ε, πλαίσιο, τις συμφωνίες, τοπικές συμφωνίες ε, που συνδέονται βέβαια με τα ρυθμιστικά κεφάλαια που παρουσιάζονται και βέβαια με τους διάφορους επιμέρους τομείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικές βέβαια οι δημόσιες προμήθειες και υπηρεσίες, αλλά αυτό που βλέπετε εδώ είναι το, ο πυρήνας της συμφωνίας και είναι σημαντικό πιστεύω. Και βλέπετε επίσης στο κάτω μέρος της διαφάνειας, 56% των των οικονομικών ε, κερδών από την TIP θα έχει να κάνει με το περιορισμό των θημερών συμφωνιών. με τον περιορισμό των εμποδίων. Άρα λοιπόν ε, θα το δούμε και αυτό. Τι είναι τα τεχνικά εμπόδια στις υπροσκόμματα συναλλαγές. Βλέπετε εδώ τα κάτω τμήματα που είναι κομμάτι και των ρυθμιστικών εμποδίων και των μη δασμολογικών φραγμών. Ρυθμίσεις λοιπόν, προδιαγραφές πρότυπα και ε, αξιολόγηση. Πρέπει να αντιμετωπιστούν λοιπόν αυτοί οι φραγμοί, αυτά τα εμπόδια. Μεγάλο κομμάτι έχει γίνει, υπάρχει βέβαια αυτή η μεγάλη σύνοδος της Μαδρίτης. Ο Πίτερ Τσέις και ο υποφαινόμενος ε, δημοσιεύσαμε στο ΣΕΠΣ ένα, μια μελέτη που ονομάζεται This Time It's Different, ε, είναι διαφορετικά αυτή φορά ρυθμιστική συνεργασία στην TTIP, πρόσφατα με τέσσερις σελίδες παράρτημα, όπου καταγράφονται οι ιστοσελίδες επί 20 χρόνια κάθε επιτεύγματος της συνεργασίας αυτής στον τομέα, με επιπλέον μια άλλη ιστοσελίδα με 72 σελίδες που παρουσιάζει όλα αυτά, τα θέματα σε λεπτομέρεια. Δεν, και αυτό το κάνω Εν, εν ολίγης, δηλαδή αυτή η δουλειά δεν έχει γίνει συστηματικά. Και οι συμφωνίες αυτές για την ε, αποδιάρθρωση των ε, μη δεσμολογικών εμποδιών, τεχνικών εμποδιών, είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να δώσει λύσεις, ό,τι και να λένε οι ε, εμπλεκόμενοι φορείς, πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Ουσιαστικά πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια προσέγγιση φιλόδοξη, με επιδίωξη των κερδών φυσικά που έχει ορίσει, αλλά και να είναι μια ζώσα συμφωνία όπως υπόθηκε νωρίτερα. Και να υπάρχουν, σοβαρά κενά. Έχουμε επίσης όμως ένα αμυντικό συμφέρον ε, για το θέμα της μία μηδέα αναγνώρισης των προδιαγραφών. Θα επισέλθω σε λίγο σε αυτό. Ναι, βεβαίως είναι ε, σχετικά ανεπαρκής η διατύπωση του κεφαλαίου του σχετικού με, τις, ε, με, τους, ε, με τα τεχνικά εμπόδια, τεχνικά εμπόδια και θα δείτε επίσης ότι Υπάρχει το κεφάλαιο κόρους, υπάρχει όμως και το, συντς, το κεφάλαιο συντς, το οποίο μπορεί να είναι κάπως πιο φιλόδοξο, αλλά αντίστοιχα στην ΣΕΤΑ έχουμε το κεφάλαιο 27, πρωτόκολλο για την αξιολόγηση της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων, το οποίο έχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Είναι μια πολύ θετική έκπληξη, λοιπόν, και άρα θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αυτόν τον δρόμο, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Τέσσερις επιλογές. Εναρμόνιση τεχνικών ε, ρυθμίσεων, εναρμόνιση τεχνικών προδιαγραφών ή προτύπων, αμοιβαία αναγνώριση τεχνικών ρυθμίσεων ή ισοδύναμα. Και χαίρομαι που το έθιξαν οι συνάδελφοι μόλις τώρα και αμοιβή γνώση προτύπων ή προδιαγραφών. Λίγες από τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών αναφέρονται σε εναρμόνιση ε, τεχνικών προτύπων. Ούτε κάνει η, ΝΑΦΤΑ, ούτε κάνει η, ε, βορειοατλαντική, η βορειοαμερικανική δηλαδή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου δεν το καλύπτει αυτό. Μόνο σε μεταφορές σε ένα πολύ περιορισμένο βαθμό. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, χωρί όμω ε, και να είναι υποχρεωτικό να περιμένουμε πάρα πολλέ εξελίξει, υπερβολικά πολλέ εξελίξει. Επί παραδείγματι υπάρχουν κάποιε διεθνεί συμφωνίε που μπορούν να οδηγήσουν σε, πιο θελοντική βάση σε εναρμόνιση, διεθνεί συμφωνίε. Εάν θέλετε θα επισέλθω σε περισσότερε λεπτομέρειε μετά. Η δε μελέτη μα ε, που κάναμε με το, μαζί με τον Πίτερ Chase ε, και μπορείτε να τη λάβετε αν θέλετε να τη διαβάσετε, αναφέρεται σε κάποιες δυνατότητες, αλλά οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Εναρμόνιση λοιπόν. Η εναρμόνιση έχει σημεία Α και Β. Μιλάει για συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και αμερικανικών υπηρεσιών προτύπων για εναρμονισμένα πρότυπα. Καλύτερα μεταξύ μιας διασύνδεσης του συστήματος ISO και ES, EEC, που είναι πιο δύσκολο να δεχθούν οι Αμερικανοί. Οπότε τίθεται το ερώτημα ποιο τελικά θα πρέπει να προχωρήσει τη συνεργασία. Γιατί θα θυμάστε ότι η Ελένα Σαντιάγο το Φεβρουάριο και ξέρετε ότι είναι γενική γραμματέα τη Ένα ΕΝΕΛΕΚ, η Λένα Σαντιάγο, μια καταπληκτική κυρία, πολύ αγωνιστική για να προσπίσετε τα συμφέροντά μα κτλ. Αλλά όταν ένα από του ε, ευρωβουλευτέ εδώ τη ρώτησε, γιατί καθόταν δίπλα μου, τι κάνετε εσείς εντωμεταξύ για να προχωρήσετε ύστερα από 25 χρόνια στην ήπια ρύθμιση του θέματο των προτύπων, Μπόρεσε να προσφέρει μόνο ένα παράδειγμα. Αυτό ακριβώ είναι το πρόβλημα. Το, το πρόβλημα είναι ακριβώ ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη όρεξη να το κάνουμε αυτό. Και ένα λόγο είναι αυτό που βλέπετε τα μικρά μικρά γράμματα να περιγράφουν. Γιατί η γενική τάση στην Ευρώπη είναι τι θα συνεργαστούμε με την ΑΝΣΥ, με την Αμερικανική δηλαδή υπηρεσία. Και όσο πιο πολύ το κάνουμε αυτό τώρα και έγινε μεγάλη συζήτηση στη Δανία με πάρα πολλούς τοποθετήσεις, τόσο και λιγότερο πιστεύουμε στην ιδέα ότι η Άνση θα είναι ο φορέα με τον οποίο θα πρέπει να διαπραγματευτούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι φορεί που παράγουν διεθνή πρότυπα, όχι όμω ISO, IEC. Πρότυπα ISDM, παραδείγματι, που χρησιμοποιούνται σε 100 διαφορετικέ αγορέ. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε απευθεία συνεργασία με κάποιου από αυτού, εκτό του πλαισίου Άνζη ή έστω με κάποια ήπια συμμετοχή τους και επίσης οι συμφωνίες ε, της Βιέννης για τα πρότυπα Βιέννης Δρέσδης ε, δίνουν ε, την ταυτόχρονη, οδηγούν σε μια ταυτόχρονη υιοθέτηση προτύπων από την ίσο την ίση. Αυτό αν το καταφέρουμε θα ήταν πολύ σπουδαία υπόθεση. Αμοιβαία αναγνώριση δεν φαίνεται να είναι τόσο καλή ιδέα γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ζητήματα της εσωτερικής αγοράς, της ελεύθερης διακίνησης που δεν θα επιτρέπουν την ε, ανάπτυξη δραστηριότητα από το δικαστήριο, άρα δεν καλύπτεται η TTIP. Ωστόσο, θα ήθελα να σας πω πώς μπορούν τα ισοδύναμα, για να δούμε τη διαφορά με την αμοιβαία αναγνώριση και τα ισοδύναμα, ή την αναγνώριση ισοδυναμίας στη συνέχεια. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι έχουμε βάλει πάνω σε, στην πάνω πάνω γραμμή ένα don't, αν θα είναι δηλαδή απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερο σε μηδέα αναγνώριση. Κοιτάξτε, όταν έχουμε τόσες προδιαγραφές στις ΗΠΑ που ισχύουν σε όλο τον κόσμο, το ISTM παραδείγματι, παρότι δεν υπάρχει αυτόματη αναγνώριση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σχέση με αυτό, είναι κατά 40% ενσωματωμένε στην παραγωγή μα Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εάν λέμε ότι δεν αναγνωρίζει τις ε, προδιαγραφές ISO, IEC, ε, το κράτο των ΗΠΑ. Εδώ έχουμε να κάνουμε, είναι γιατί έχουμε να κάνουμε μια πρακτική αναγνώριση των δικών του προτύπων σε 40-60 χρόνια σε όλο τον κόσμο και δι' όλη την Ευρώπη. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιμένουμε ότι πρέπει να περάσουν στο ISO ή εσύ. Γιατί υπάρχει κάτι που έχουν επικυρώσει με τη συμπεριφορά τους οι αγορές και οι, Αμερικανοί, και οι ε, παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε μια λύση. Χωρίς να επιμένουμε σε δογματικά ζητήματα βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα ναι πρέπει να επιμένουμε σε η ζωή σε μακροπρόθεσμα αλλά όχι βραχυπρόθεσμα. Και επίσης πρέπει να στήσουμε από πλευράς Αμερικανών και εμείς περισσότερη ευελιξία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ένα από τα πιο σοβαρά πράγματα για τον τρόπο, τα πιο σημαντικά είναι για, για τον τρόπο με τον οποίο περνάνε οι δικές μας οι προδιαγραφές στο Αμερικανικό Δίκαιο είναι η περίφημη εγκύκλος Α119. Και άρα αυτό μπορούμε να το διασυνδέσουμε με την TTIP για να δώσουμε λύση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μέσω αυτού. Διάφορες λοιπόν επιλογές που μπορεί να προβάλλει η ευρωπαϊκή πλευρά για να απαιτήσει πράγματα από την αμερικανική και επίσης λύσεις για να ικανοποιήσουμε αιτήματα των Αμερικανών. Δεν έχω όμως τόσο χρόνο και γι' αυτό θα περιμένω τα ερωτήματά σας για να δώσω σχετικά απαντήσεις. Στην αξιολόγηση προσαρμογής πάλι έχουμε ένα ζήτημα. Έχουμε μακροπρόθεσμα, μακροχρόνιο μάλλον με την... ε, ε με την ηλεκτρομηχανική και τα ηλεκτρικά γενικά, με την όσα όπως ονομάζεται που είναι η σχετική υπηρεσία των ΗΠΑ, που κάνει πολλά πράγματα, αλλά θα πρέπει να αλλάξουν και πολλά πράγματα υπέρ των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ενημέρωση για την ε, μηχανική και, τους, ε, και τις μηχανές, όπου υπάρχουν λύσεις μεταξύ τριών επιλογών για τις υπηρεσίες αξιολόγησης προσαρμογής στα πρότυπα, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα γίνει, τεράστια προβλήματα λοιπόν για τον ανταγωνισμό. Δεύτερο, να μην επαναλαμβάνονται οι δοκιμές των συστατικών, που πολλές φορές δοκιμάζονται πριν να μπουν μέσα στη μηχανή και μετά ξαναδοκιμάζονται να μπουν πάνω στο μηχάνημα, κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να γίνεται. Αυτό επιβάλλει πάντα η UL, που έχει τεράστια και κυρίαρχη θέση στην Αμερικανική αγορά. Και τρίτον, πρέπει να επιβάλλουμε μια πειθαρχία στη UL και να συγκρατήσουμε αυτή την κυριαρχική της θέση και στάση. Μετά που έχει συνέπεια τεράστιες αυξήσεις τιμών για προϊόντα που προξενούνται από τι τάσει τη. Ακόμα καλύτερο όμω είναι να δούμε το παράδειγμα της ε, ΣΥΤΑ με το MRA, το οποίο χάρη στην αμοιβαία αναγνώριση έδωσε λίστα προβλήματα. MRA συμφωνία έχουμε με τις ΗΠΑ και πρέπει να, το, να την επεκτείνουμε τη συμφωνία αυτή ώστε να καλύψει και άλλους τομείς. Φερρυπίν, ιατρικά μηχανήματα όπως και στη ΣΕΤΑ που είναι πολύ πιο ανοιχτός πλέον ο τομέας από όταν είναι πριν. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ε, να περιμένουμε πάρα πολλές ε, επιτυχίες. Ε, με την Αναμπέλα Κορέα κάναμε μια μελέτη το 1989 όπου καταλήγουμε ότι από τους τρεις εκ των έξι τομέων όπου απέτυχε η τυποποίηση, η, η, η μορφής ρυθμιστική προσαρμογή είχε καλύτερα αποτελέσματα από την επιβολή κανόνων, δηλαδή με εθελοντικούς κανόνες, φερρυπίν στα ιατρικά, είτε μηχανήματα είτε προϊόντα, φάρμακα. Μπορούν να υιοθετούνται κανόνες ή πρότυπα ρυθμιστικά επαναλαμβάνω, από τις αρχές δηλαδή οι οποίες ε, η μία εμπιστεύεται την άλλη, από αντίστοιχα κράτη, Υιοθετούν λοιπόν του ίδιου κανόνε σε μια σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ του, οι οποίοι κάνουν ισχύουν για την εσωτερική αγορά και έτσι, και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το καταφέρει η TTIP, μπορούμε να έχουμε κατευθυντήριε γραμμέ ταυτόσιμε. Η δε μείωση του κόστου στην, ε, για τα προϊόντα αυτά είναι πολύ σημαντική. Η ρυθμιστική λοιπόν συνεργασία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και για να καταλήξω, πριν σας εκφράσω και τι ευχαριστίε μου, ε, θα ήθελα να δώσω κάποιες πιο συγκεκριμένες προτάσεις και ιδέες. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες πρέπει να προχωρήσουν περισσότερο προς τις προδιαγραφές ISO ESE. Αυτό όμως πρέπει ταυτόχρονα να συμπεριλάβει και την ιδέα ότι έχουν τεράστια αποδοχή στις αγορές εδώ και δεκαετίες οι εννέα μεγάλες ρυθμιστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο και την Ευρώπη και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τους επιτρέψουμε να ενταχθούν στο, στην συμφωνία και μακροπρόθεσμα να μπουν στο σύστημα ISO ESE. Παράδειγμα, όταν κατασκευάζεται ένα αεροπλάνο, η ΆΤΑ, η ΆΣΑ θα πρέπει να δώσει την πιστοποίηση ασφάλειας. Ε, εκεί χρησιμοποιεί τις προαμερικανικές προδιαγραφές, ISM τις οποίες επίσης χρησιμοποιούν πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες. Δεν είναι απλώς ISTM δηλαδή οι προδιαγραφές αυτές. Υπάρχει μια αμερικανική Ευρω... και ευρωπαϊκή μαζί υπηρεσία που μελετάει τις προδιαγραφές των συστατικών, των ε, εξαρτημάτων και μπορούν ως εκ τούτου εξυπηρετώντας τις ανάγκες και ευρωπαϊκών και αμερικανικών επιχειρήσεων να συμφωνήσουν πάνω σε αυτά τα πρότυπα. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε και την άλλη πλευρά. Και επιπλέον σε σχέση με τις ε, προδιαγραφές οι οποίες έχουν ενταχθεί στην νομοθεσία στις πολιτείες. Ε, εκ των αυτών κυρίων φορέων πιστοποίησης, οι μισές τουλάχιστον καλύπτονται νομοθετικά. Άρα πρέπει να στραφούμε και σε αυτές. Είναι συνομιλητής μας, για αν θέλουμε επιτυχία. Και κλείνω λέγοντας ότι χρειάζεται και τις προδιαγραφές και την αξιολόγηση της προσαρμογής να αντιμετωπίσουμε από κοινού και επίσης πρέπει η Ευρώπη να δεχθεί ότι υπάρχουν πολλοί τομείς αυτοδήλωσης σε αυτό που ονομάζεται τώρα ρυθμιστικό πλαίσιο και οι Αμερικανοί σε αυτούς τους τομείς και δεν είναι λίγοι μπορούν να ενταχθούν με αυτοδήλωση με self-declaration, ενώ εμεί ως Ευρωπαίοι δεν μπορούμε να το κάνουμε στην Αμερικανική αγορά. Το 2008 λοιπόν αυτό που συνέβη ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στην όσα μια αριθμιστική αρχή αμερικανική, να έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να μπαίνουμε με το self-declaration στην αμερικανική αγορά. Ύστερα από δύο χρόνια ερευνών, έγινε μια εξαιρετικά λεπτομερή μελέτη συνεπειών και αξιολόγηση κινδύνου, με όλες τις δυνατές δοκιμές και δοκιμασίες και ελέγχους, με αποτέλεσμα ότι η ΩΣΑ δεν δεχόταν αυτή την αυτοδήλωση, διότι υπήρχαν ελλείψεις ανεπάρκειες στο σύστημα του self-declaration το ευρωπαϊκό και την αγορά μας και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, διότι αν δεν είχαμε αυτό, τα κενά, αυτές τις αδυναμίες στο σύστημα μας, οι Αμερικανοί θα τα είχαν δεχτεί. Θα είχαν δεχτεί να κάνουμε κι εμείς self-declaration. Με πολύ χαμηλότερο κόστος λοιπόν από τα προκαλούμενο από τα τεχνικά εμπόδια στο χώρο της μηχανικής και των μηχανημάτων. Και πρέπει να κοιτάξουμε το γεγονός ότι αυτές οι εξαγωγές είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι αντιστοιχεί στι εξαγωγέ τη αυτοκινητοβιομηχανίας και της χημικής βιομηχανίας μαζί προ τι ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έφτασαν και τρει βασικοί διαπραγματευτέ τη Κομισιόν. Μπορείτε να σηκώσετε λίγο τα χέρια σα να σα δουν οι παριστάμενοι. Λίνα Λουελέη, Φερνάντο Πάροτ ε, για τους δασμούς και Παύλο Νέρα για τα πρότυπα. Οπότε μπορούν να απαντήσουν και οι ίδιοι σε ερωτήσεις. Πριν ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις, ε, θα πω το εξή. Ε, δεν ξέρω ποιες είναι οι εμπειρίες σας, αλλά εγώ έχω πάρει 7.000 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φτάνουν και άλλα. Θέλω λοιπόν να στείλω σε όλους αυτούς ε, εξηγήσει ε, με επιχειρήματα σε μια γλώσσα την οποία να την καταλαβαίνουν. Οπότε, αν είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιούμε ιδιόλεκτο ε, ακρόνημα κλπ. Θέλουμε να τα χρησιμοποιούμε, να τα χρησιμοποιούμε πολύ προσεκτικά και με φιδό. Ε, ακόμα και στις ε, ε, παρουσιάσεις που είδαμε υπήρχε ένα ακρόνημα το οποίο ο εμπειρογνώμονάς μου δεν κατάλαβε. Οπότε παρακαλώ πολύ να προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε σαφή γλώσσα για να βοηθήσουμε και του υπόλοιπου. Ο κ. Φάμπ ήταν ο πρώτος ομιλητή δεν είναι εδώ. Εύλιν Γκέφχαρτ. Πρώτη ερώτηση. Και μετά θα περάσουμε στι υπόλοιπε ομάδε. Ναι, ευχαριστώ. Με καλύψατε ω προ την πρώτη μου παρατήρηση. Και εμεί θέλουμε με τη σημερινή μα συζήτηση, και η οποία διαβιβάζεται μέσω του διαδικτύου και, και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να την παρακολουθούν. Θέλουμε λοιπόν και εμείς να έχουμε μια γλώσσα που θα μπορεί να καταλάβει ο μέσος πολίτης. Οι πολλές λοιπόν ε, τα πολλά ακρονίμια και μάλιστα όταν ο μιλητής δεν, δεν έχει μητρική γλώσσα την αγγλική και άρα έχει ζήτημα και στην προφορά του, δεν μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε με τόση ευχέρεια την ομιλία του, πράγμα το οποίο είναι λυπηρό διότι χάνεται αρκετή πληροφορία. Και θα ήθελα Ξέρω ότι είναι δύσκολο για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται τόσο εντατικά και σε βάθος με την υπόθεση αυτή, αλλά θα ήθελα να γίνει μια προσπάθεια, ώστε να μπορούν όλοι να καταλάβουν. Πολλές είναι οι ερωτήσεις μου. Θα αναγκαστεί να κάνω μια διαλογή, γιατί διαφορετικά δεν θα αφήσω χρόνο για τους υπόλοιπους. Αν και πρέπει να πω ότι όσο πιο πολλά μαθαίνω, τόσο πιο πολλές ερωτήσεις μου γεννώνται. Με ενδιαφέρον λοιπόν να ακούω αυτό που ο κύριος Μπέρκμανς, ότι η αμοιβαία αναγνώριση δεν πρέπει να υιοθετηθεί. Χαίρομαι ιδιαίτερος, διότι έτσι αποφεύγουμε και άλλες σχετικές δυσκολίες, τις οποίες έχουμε άλλωστε καλύψει μια συζήτηση σχετική με την παροχή υπηρεσιών. Εάν η αρχή της προελε... χώρας προελεύσεως πρέπει να διατηρηθεί ή όχι. Και γι' αυτό και νομίζω ότι η έννοια της ισοτιμίας είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε κάποιες πιο λεπτομερείς ιδέες για το πώς μπορεί να εκφραστεί αυτή η έννοια της ισοτιμίας, τι εννοείται ακριβώς, ή αν θέλετε να μας δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις σκέψεις σας. Κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι, και με συγχωρείτε τη λησμόνισα τα ονόματά σας, δεν τα βλέπω στο πρόγραμμα, στη ρυθμιστική συνεργασία και την ισοτιμία. Λέγεται ότι θα βελτιωθεί το επίπεδο των προτύπων Θέλω πολύ να το πιστέψω αυτό, αλλά δώστε μου μερικά παραδείγματα, ή επιχειρήματα, πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Γιατί πολλά από τα μηνύματα, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που μου αποστέλλονται, αναφέρονται ακριβώς σε ανησυχίες για μείωση του επίπεδου των προτύπων. Και θέλω και εγώ να έχω επιχειρήματα για να απαντήσω σε αυτό. Πώς θα το καταφέρουμε στα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα, Φερρυπίν. Έχουμε τεράστιες διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, Ηνωμένων Πολιτειών ως προς τις προϋποθέσεις ασφαλείας, ποιότητας καλύτερα. Τι θα γίνει λοιπόν. Τρίτο δε και τελευταίο ερώτημα από πλευράς μου, εκ των πολλών που είχα να καταθέσω, δημόσιες προμηθείς. Λέτε ότι έχουμε ευρωπαϊκέ ρυθμίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει η ιστορική αγορά, όλοι έχουν να αντιμετωπίσουν τι ίδιε ρυθμίσει. Αυτό όμω δεν ισχύει στι ΗΠΑ γιατί κάθε πολιτεία έχει διαφορετική ρύθμιση. Έστω. Αλλά μπορεί να ισχύει, αλλά όχι πλήρω, διότι το ευρωπαϊκό δίκαιο έχει και πολλέ διατάξει για τις οποίες αναφέρεται ότι στις δημόσιες προμήθειες η εξαγωγή ε, της διαδικασίας θα οριστεί σε σχέση με ορισμένα στοιχεία από τις κρατικές αρχές για το πώς προτιμούν να διεξαγάγουν αυτήν την ε, διαδικασία. Και πολλές είναι οι φορές όπου θερυπίνει για τη Γερμανία αναφέρεται πως κάποια κριτήρια, αναφέρεται από την νομοθεσία, πως κάποια κριτήρια ε, ε πόκινται στην διακριτική ευχέρεια των ομοσπονδιακών κρατηδίων για το αν θα εφαρμοστούν ή όχι. Άρα δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη ομοιομορφία και δεν έχουμε να κάνουμε κριτήρια που έχουν να κάνουν και με την ποιότητα, έχουν να κάνουν και με την προέλευση. Και με τις προϋποθέσεις, φερειπίν, ε, τήρηση συλλογικών, όρων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πολλά εξαρτώνται από αυτές τις διατάξεις. Όταν λοιπόν λέμε ότι ε, καταλύουμε φραγμούς, δεν πρέπει αυτό να σημαίνει ότι θα καταληθούν και οι φραγμοί τους οποίους εμείς έχουμε ορίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εχέγγυα ποιότητας. Η ε, Πρόεδρος. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω το ρολόι από ένα λεπτό ο καθένας. Λυπάμαι πολύ εύληνα, αλλά δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε απαντήσεις από τους εμπειρογνωμονές μας. Ο Ανδρέας Σφάπ έχει το λόγο. Ναι, Πρόεδρε. Για να δώσω μια, έναν αντίλογο στα είπε η κυρία Γκέπχαρτ. Βεβαίως και δεν έχει πάρα πολλά περιθώρια το εθνικό κράτος να εμπλακεί στο ζήτημα της διαμόρφωσης των τοπικών διατάξεων για τις προμήθειες. Θα ήταν ε, αντίθετο με το ευρωπαϊκό δίκαιο το να υπάρξει κάτι τέτοιο, ενώ στο αμερικανικό δίκαιο έχει πολύ σημαντικό μερίδιο των ε, προμηθειών το επίπεδο, το τοπικό ή το πολιτιακό. Είναι μεγάλο το ποσοστό δηλαδή επί του ΑΕΠ. Και θέλω να ρωτήσω του ομιλητέ μα εδώ ή τον ομιλητή μα καλύτερα. Μπορούμε να αναμένουμε ότι σε επίπεδο ομοσπονδιακό ε, επίπεδο στι ΗΠΑ θα έχουμε σύντομα ή κάποια στιγμή σε μια δεκαετία ε, την ανάληψη τέτοιου είδους συμβάσεων θα έχει αναχθεί δηλαδή από το πολιτιακό στο κρατικό επίπεδο αυτή, το σύνολο αυτών των διαδικασιών για τις δημόσιες προμήθειες ή θα παραμείνει πάντα στο πολιτιακό επίπεδο. Θα έχω πολλές ερωτήσεις, θα είμαι σύντομος όμως. Σε ό,τι αφορά τις κρατικές ε, προμήθειες, δημόσιες συμβάσεις, ε, πώς θα τους πείθετε να δεχτούν τις προτάσεις μας τι μπορούμε να τους πουλήσουμε και πώς μπορούμε να τους το πουλήσουμε για να το δεχτούν. Επίσης, μιλάμε για ελεύθερη ε, για ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Αν δείτε το Buy America, ε, προωθεί την ε, τοπική εγκατάσταση μεγάλων εταιριών για να έχουν πρόσβαση στην αγορά. Αυτό όμως ε, δεν βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Μετά, δεσμοί. Δασμοί. Ε, είπατε ότι εκεί έχουμε μικρή δυνατότητα βελτίωση. Αν δείτε όμω τη διαφορά στι τιμέ καταναλωτή ανάμεσα στι ΗΠΑ και την, Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, είναι τεράστιε διαφορέ. Ε, iPhone για παράδειγμα είναι 150 ε, δολάρια πιο φτηνά εδώ από, ε, πιο ακριβά εδώ από τις ΗΠΑ. Ε, ε, άρα λοιπόν θα είχαμε πολύ μεγάλο όφελος αν μειώναμε τους δασμούς. Ευχαριστώ. Δίτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ όλους όσους με έκαναν παρουσιάσεις και για το ε, περιεχόμενο και για τον ενθουσιασμό τους. Χαίρομαι που ε, μου επιβεβαιώσατε ότι η γνώμη μας και η γνωμοδότησή μας ήταν σωστή. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, ε, βασική προτεραιότητα συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης χαίρομαι που καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία GPA ε, ε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, δεν είναι αρκετή. Ε, η συμφωνία για να προτιμήσεων δηλαδή δεν είναι αρκετή. Ε, τι θα χρειαστεί, ποιο επιχείρημα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να πείσουμε τους, τους Αμερικανούς να, να μπουν σε αυτή τη συμφωνία και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως, ως βουλευτές για παράδειγμα να διοργανώσουμε μια συνάντηση με τις ενώσεις των κυβερνητών ε, έτσι ώστε να καταλάβουν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τους φραγμούς, δασμολογικούς και μη δασμολογικούς, ε, χαίρομαι για τα συμπεράσματά σας, τα καλωσορίζω. Ε, προφανώς υπάρχει ε, ένα όφελος το οποίο αναμένουμε από την απόσυρση των την κατάργηση των φραγμών. Ε, επίσης ο διάλογος μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών πολύ σημαντικός, ε, ε ρυθμιστική συμφωνία ε, και το γεγονός ότι θα είναι μια ζώσα συμφωνία είναι πολύ καλό. Επίσης να ζητήσω από την Πρόεδρο, δεδομένου ότι η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και έχουμε τόσα πολλά ζητήματα, να θίξουμε. Μήπως θα μπορούσαμε να την επαναλάβουμε. Πρόεδρος, παρακαλώ, αν μπορούμε να περιστούμε σε ερωτήσεις μόνο. Δεν θέλω να διακόψω τη συζήτηση ε, ή θέλουμε να κάνουμε συζήτηση. Θα ε, επανέλθω σε σένα αν έχεις κάποιες πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δεν Δεν είναι εδώ. Πασκάλ. Ε, ε. πολύ γρήγορα, Βίκη γιατί πρέπει να περιοριστούμε σε ερωτήσεις. Εγώ όμως δεν έχω να θέσω ερωτήσεις, απλά να πω. Ε, η Ντίτα μόλις μίλησε για τον ενθουσιασμό. Όταν ο ενθουσιασμός πλησιάζει την προπαγάνδα, εγώ ανησυχώ. Δεν θέλω λοιπόν να κάνω ερωτήσεις. Θα αρκεστώ στο να κρατήσω, να διατηρήσω τη δική μου γνώμη του θέματος. Θα έχετε χρόνο για απόψεις. Αυτή τη στιγμή θέλω να περιοριστούμε σε ερωτήσει. Ε, Φιλίπ Ζουβά. Ναι, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, αν δούμε τα νούμερα της Κομισιόν, στην πραγματικότητα, είπα, ε, ε, εφαρμόζουν προστατευτισμό στις δημόσιες συμβάσεις. Είπαμε το 30% μόνο ε, των αγώνων στην Αμερική είναι ανοιχτέ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη 80%. Έτσι ορίζεται για μας ο προστατευτισμός και θέλουμε να δούμε κατά πόσο εμπειρογνώμονες επιβεβαιώνουν αυτά τα νούμερα. Δεύτερον, ήθελα να πω ότι και τα δύο μέρη ε, ψηφίζουν υπέρ διαφάνεια, της διαφάνειας. Ε, ακούω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας στέλνει ε, κάποια ενημέρωση γραπτά ότι τα νούμερα που δίνουν οι Αμερικανοί είναι του 2008 και από το 2008 και μετά δεν υπάρχουν ε, πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα των αγορών. Θέλω να μου το επιβεβαιώσουν εμπειρογνώμονε. Τρίτον, μου λένε ότι οι ΙΠΑ θέλουν να ανοιχτούν, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να εξοπλιστούν με επιπλέον νομοθεσία που εφαρμόζει ε, προστατευτισμό. σκεφτούμε την πράξη Buy America, θέλω να μου πούνε οι ειδικοί τι σκέφτονται και μετά για την Κομισιόν με καθησυχάζει ε, η κόκκινη γραμμή που αναφέρατε αυτή η τεράστια συμμετρία των δημοσίων συμβάσεων όμως ε, ανησυχώ και επαρθύνομαι στην Κομισιόν βάσει μια απάντηση που μου έστειλαν πρόσφατα μου εξήγησαν ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να αυξήσουν το άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων σε 85 έως 95% στα, στα κράτη-μέρη της MP. Ε, ε, ε, εγώ δεν σας κρύβω ότι θέλω να υπογραφεί η σύμβαση αυτή, αλλά όσο ακούω τα νούμερα τόσο περισσότερο ανησυχώ. Ελπίζω να αλλάξω γνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ανά Μαρία. Ευχαριστώ. Πριν μπούμε στο τεχνικό ερώτημα, υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα από ό,τι βλέπω διότι επιτέλους συζητάμε τα πράγματα όπως έχουν βλέπουμε ότι το μοτίβο που προκύπτει, ε, αυτό που επαναλαμβάνεται συνεχώς, είναι η έλλειψη πρόοδο από πλευράς ΙΠΑ, ο κατεκριματισμός του συστήματός τους, η απροθυμία τους να προχωρήσουν σε ε, γενικά πρότυπα, καθολικά, παγκόσμια και σε ρυθμιστική σύγκληση στις δημοσίες συμβάσεις. Το θέμα ουσιαστικά είναι πώς θα ενισχύσουμε τις διαπραγματικές μας εξουσίες αντί να βάζουμε κόκκινες γραμμές στην Κομισιόν. Εγώ ήθελα να μάθω περισσότερο από εσάς, όπως είπε και η Εύελεν, αν όχι αμοιβαία αναγνώριση, αφού λέτε ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την οδό, τι τότε. Ποια θα μπορούσε να είναι η συνεργασία μεταξύ οργανισμών τυποποίηση, πώ θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό στο μέλλον, να καθίσει ο τομέα τη βιομηχανία, ε, και από των δύο πλευρών και να συζητήσει κοινά πρότυπα για το μέλλον. Ποιοι τομεί πιστεύετε από τεχνική άποψη θα μπορούσαν να σημειώσουν κάποια ε, πρόοδο. Αλλά η ερώτηση κλειδί είναι πώ θα καλύψουμε το χάσμα μεταξύ των όσων λέτε εσεί που είναι οι πραγματικέ προκλήσει και τη δημόσια συζήτηση που είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Ε, λέτε σαφώ ότι η νομοθετική εθνική κυριαρχία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοινοβουλίου ε, βρίσκεται σε κίνδυνο. Αλλά εμείς είδαμε αυτή την ομοφωνία στην Ολομελία ε, την περασμένη εβδομάδα και ζητώ συγγνώμη Βίκη, αλλά εκεί τα πράγματα κατέρευσαν. Όταν έχουμε μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες που έχουν συμφωνήσει στην Επιτροπή και μετά στην Ολομέλεια δεν ακολουθούν αυτό που είπαν και δεν έχουμε προλάβει να το συζητήσουμε Θέλω να μας βοηθήσετε να καλύψουμε αυτό το κενό. Και παρακαλώ μην μου λέτε από την μια μεριά όσα ε, στη μια διαφάνεια και την ποιτή στην άλλη. Ξέρετε, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν αυτή τη γλώσσα. Όλα αυτά τα κρονίμια δεν τα αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτε. Λοιπόν, να σα ε, πω ποιου έχω στον κατάλογο μιλητών. Πρώτα έχω, πρώτα έχω τον Νίκολα Ντάντε, τη Λίσα Γιακονσάρη, Γετς Νίλσεν και μετά και μετά θα επανέλθουμε στο ένα διότι προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήσεις ε, και ελπίζουμε να, να έχουμε αρκετό χρόνο να περάσουμε και στην επόμενη συζήτηση. Λοιπόν, Νίκολα, λοιπόν, έχω να πω πρώτον, όπως είπαμε πολλές φορές, σε πολλές συναντήσεις, δεν θέλουμε να χαμηλώσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δεύτερον, θέλουμε να είναι φιλόδοξη η TTIP. Τρίτον, αυτό που συζητάμε σήμερα, δηλαδή η ρυθμιστική σύγκληση, θα πρέπει να αποτελέσει το σημαντικότερο κομμάτι της TTIP που θα αποφέρει περισσότερο περισσότερα ωφέλη εγώ τώρα τα νούμερα δεν τα πολύ πιστεύω, 55% κέρδη και όλα αυτά. Τα νούμερα αυτά αλλάζουν ανάλογα με το ποιο τα δίνει. Αλλά ανεξάρτητα από τα ποσοστά, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ θετικά από οικονομική άποψη. Και μετά ε, κυρίω μπορούν να δώσουν πολλέ ευκαιρίε στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Πέραν όλων αυτών, όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια εμπορική συμφωνία σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιλύσουμε όλα τα αριθμιστικά ζητήματα. Ε, ούτε καν μέσα στην επόμενη δεκαετία ε, ε, ακόμη και αν διακούσαν οι διαπραγματεύσεις 10 χρόνια. Εγώ θέλω να ρωτήσω με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία προοδευτικά θα επιχειρεί να καταστήσει ομοιόμορφα τα πρότυπα ώστε να υπάρχει μια ρυθμιστική συνεργασία, μια ρυθμιστική ομοιομορφία για να συνεχίσουμε με στα επόμενα χρόνια, διότι το κεντρικό ερώτημα είναι τι ακριβώς εντός της συμφωνίας θα μπορούσαμε να ε, ορίσουμε εμείς ως μέθοδο, όχι συμφωνία επί των πάντων, διότι σίγουρα θα μπορέσει να υπάρξει κάποια συμφωνία εύκολα για κάποια θέματα, ενώ για άλλα θέματα όπως η ρυθμιστική συνεργασία, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Οπότε δεν μπορούμε να, αναμένουμε ότι θα βρούμε συμφωνία σε όλα τα θέματα αμέσως. Ε, ευχαριστώ. Λίσα. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε ε, η συμφωνία ε, TTIP θα αποτελέσει εξωτερικό κίνητρο, είπατε, για να αρθούν οι εθνικοί φραγμοί και αυτό φοβάται ο κόσμος. Για παράδειγμα, στον τομέα της εξόρυξης, η φραγμή αυτή οφείλεται στο γεγονό ότι η εθνική νομοθεσία λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον, οπότε εκεί το ερώτημα των προτύπων των standards. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν συζητάμε το θέμα σε εθνικό επίπεδο. Εσείς αναφέρατε τα αεροσκάφη για παράδειγμα, αυτό είναι ένα παράδειγμα φυσικά. Εκεί από όσο κατάλαβα τα πρότυπα είναι υψηλότερο επίπεδο στους είπα από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μαζί με αυτή τη συμφωνία, παράλληλα με αυτή τη συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να, να, το, να προχωρήσουμε την εθνική συζήτηση επί του θέματος. Ε, ε, λοιπόν, ναι, συμφωνώ με τον κύριο Ντάντη, ο οποίος λέει ότι όταν έχουμε μία συμφωνία θα πρέπει να έχουμε και ένα μηχανισμό όπου θα συνεργαζόμαστε για αριθμιστικά θέματα αν μη τι άλλο, για τα ε, δικαιώματα των καταναλωτών. Αλλά η ερώτηση μου, λέει ο κ. Νίλσον, οφείλεται, αφορά τις δημοσίες συμβάσεις. Όπως είπε η Εύλεν, έχουμε μια νέα οδηγία, η οποία ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά υπάρχει περιθώριο λιγμών. για παρεκκλήσεις σε περιφερειακό επίπεδο, σε κρατικό επίπεδο, ακόμη και αν υπάρχουν, είναι μικρές αυτές οι παρεκκλήσεις. Αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι η ύπαρξη διαφορετική νομοθεσία τη ΕΠΑ. Δηλαδή, όταν θα έχουμε μια συνεργασία με μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, τα πράγματα θα είναι πάλι διαφορετικά. Γιατί και αυτή η κάθε πολιτεία έχει του δικού τη κανονισμού. Αυτό διαφαίνεται ω πρόβλημα. Είναι λοιπόν διατεθειμένε οι να κάνουν κάτι γι' αυτό. Για να υπάρχει διαφάνεια και στο δικό του ε, σύστημα, ώστε η νομοθεσία να μπορεί να καλύψει όλη τη χώρα. Ευχαριστώ να αφορά όλη τη χώρα. Αφήσε ναι. ναι. Ε. Ευχαριστώ. Ε, κοιτάξτε, πολύ καιρό μας λένε ότι η συνθήκη αυτή θέλουμε να ορίσει κοινά πρότυπα. Εγώ χαίρομαι που ακούω κάτι, φανταζόμουν εδώ και καιρό ότι το ζήτημα των προτύπων δεν θα ρυθμιστεί μέσω συμφωνιών αλλά μέσω οργανισμών τυποποίησης που δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να τη συμπεριλάβουμε στο πεδίο εφαρμογή αυτή τη συμφωνία. Μετά τίθεται το ζήτημα του κόστου, των τεχνικών φραγμών, των μέτρων προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντο. Γιατί όχι, το ζήτημα του κόστου ε, σίγουρα είναι σημαντικό. Αλλά αυτά, ξέρετε, τα προστατευτικά μέτρα τα υιοθετούμε διότι προσθέτουν αξία σε κοινωνικό, σε περιβαλλοντικό επίπεδο ε, αξία που δεν πουλιέται απαραίτητα, δεν έχει τιμή απαραίτητα. Όταν η ανάλυση λοιπόν εστιάζεται κυρίως στις δαπάνες, ε, θέλω να δω πώς θα ε, απαντήσουμε στις ανυπόστατους ισχυρισμούς ότι η συνθήκη αυτή, η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει σε βελτίωση των προτύπων μας. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει οτιδήποτε, οτιδήποτε αποδεικτικό στοιχείο που να στηρίζει ε, κάτι τέτοιο. Επίσης μιλάμε για τον κατακαιρματισμό της εσωτερική αγοράς, της αμερικανικής ε, αγοράς, η οποία είναι το ίδιο κατακαιρματισμένη αν όχι περισσότερο. Ε, να δούμε τι θα γίνει με τις δημοσίες συμβάσεις, με την ασυμμετρία που ανέφερε ο Φιλίπ Ζουβά και βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να καλυφθεί αυτό το χάσμα, πώς ξέρουμε ότι δεν θα βρεθούμε στην ίδια κατάσταση και σε άλλους τομείς με αμφισβήτηση τελικά των και με τεράστιο άνοιγμα προς τις αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα η αμερικανική αγορά παραμένει σε μεγάλο βαθμό μη προσπελάσιμη για τις δικές μας επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Σεχνάλοβα. Ε, μια πολύ σύντομη ερώτηση. Ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις. Μια από τις τελευταίες διαφάνειες που μας δείξατε ε, παρουσιάζει κάποια συμπεράσματα και λέει ότι η ε, ρυθμιστική εξουσία ε, δεν θα επηρεαστεί από την TTIP. Γιατί δεν θα επηρεαστεί μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Clear ερώτηση. Ντάν. Για το θέμα ε, ε, το ρυθμιστικό. Ε, πώς μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα στους τομείς ε, όπως τα crash τα οποία δεν χρειάζεται να έχουμε διαφορετικές ε, ε, που, που, που, που δεν, μπορεί, δεν χρειάζεται να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις και αυτά στα οποία μπορεί να επιτρέψουμε διαφορετικές προσεγγίσεις όπως το θέμα των τροφίμων. Και εγώ θέλω μερικέ ερωτήσει, λέει κύριε Φόρντ. Ε, στην πρώτη σα παρουσίαση είπατε ότι οι μικρέ επιχειρήσει είναι αυτέ που πιο πολύ θα ωφεληθούν από, ε, από ε, τι αλλαγέ στι ε, δημόσιε συμβάσει. Μπορείτε να το στηρίξετε αυτό σε συγκεκριμένε ιστορικέ, σε συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα. Δεύτερον, στη δεύτερη παρουσίαση αναφέρατε ότι φαίνεται πω ε, τα πρότυπα για τους κατανοητέ. Ε, δεν θα χαμηλώσουν αλλά θα ψηλώσουν. Σε τι το στηρίζεται αυτό. Ε, Επίση, ε, σε ό,τι αφορά την τρίτη παρουσίαση, θα μπορούσατε όλα τα ακρονίμια να τα εξηγείτε σε υποσημειώσεις. Σε κάθε σελίδα. Δεύτερον, λέτε στην παρουσίασή σας το εξής. SHEC, στόχοι ε, τι σημαίνει το SHEC, ε, ότι δεν είναι θέμα. Αυτό είναι safety, health, ε, ασφάλεια, υγεία, καταναλωτέ. καταναλωτές, τι, δεν το καταλαβαίνω πολύ καλά. Επίση, το κοινό θέλει ανεξάρτητες γνώμες, ανεξάρτητες απόψεις, δεν θέλει απόψεις οι οποίες να πατρονάρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Οπότε θα ήθελα τα ονόματα των συγγραφέων να βρίσκονται πάντοτε στην πρώτη σελίδα έτσι ώστε να γίνει σαφές, να γίνεται σαφές κάθε φορά ότι την έκθεση, τη μελέτη, οτιδήποτε την συνέγρεψαν και την επεξεργάστηκαν ανεξάρτητοι μυρογνώμονες. Η Κομισιόν θέλει το λόγο επίσης νομίζω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ονομάζομαι Φερνάντο Περοντεπίνη. Είμαι συντονιστές, συντονιστής της ομάδας των διαπραγματευτών. Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν θα μειωθούν τα πρότυπα. Δεν θα μειωθούν, δεν θα χαμηλώσει ο πύχης. Το έχουμε πει αυτό. Η συνέπεια, πιο πιθανή συνέπεια, είναι η προστασία να βελτιωθεί, να γίνει πιο αυστηρή. Για γιατί το λέω αυτό. Για παράδειγμα, αμοιβαία αναγνώριση των επιθεωρήσεων των ε, εγκαταστάσεων παραγωγής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Αυτό, αυτές οι επιθεωρήσεις γίνονται μέσω ελέγχων και από φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την FDA των ΗΠΑ, την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων. Αυτή αυτές οι επιθεωρήσεις θα οδηγήσουν σε βελτίωση του συστήματός μας, των συστημάτων μας. Οι επιθεωρήσεις που γίνονται για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αν γίνουν από κοινού ε, με τις επιθεωρήσεις που γίνονται στις ΗΠΑ θα γλιτώσουμε προσωπικό και χρόνο για να το αφιερώσουμε αλλού. Επίσης, τα οχήματα, το ίδιο. Εντοπίζουμε τρεις τομείς όπου μπορεί να γίνει μια επιταχυμένη εναρμόνιση. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα ε, εργαστούμε για να κατακτήσουμε εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία προφανώς δεν θα είναι χαμηλότερα σε ό,τι αφορά την προστασία τους από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε τεχνικά, ούτε νομικά, ούτε πολιτικά θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Κανέ, καμία αριθμιστική αρχή δεν πρόκειται, δεν έχει ποτέ προτείνει, ποτέ προτείνει σε 300 ώρες διαπραγματεύσεων μείωση χαμήλωμα των προτύπων της προστασίας. Δεν υπάρχει πουθενά καμία ένδειξη για το ότι υπάρχει περίπτωση να χαμηλώσει ο πύχης. Συμφωνούμε πλήρως με τα συμπεράσματα της έκθεσης που είδαμε σήμερα και με αυτήν του κ. Πέκμαντς και αυτήν που αφορούσε την προστασία των καταναλωτών. Γιατί αυτές οι εκθέσεις βασίζονται σε δεδομένα, είναι τεκμηριωμένες. Και έτσι πρέπει να εργαστούμε, όχι με βάση ισχυρισμούς. Τελευταία κάποιοι λένε ότι το e-labeling ε, μπορεί να αντικαταστήσει ε, ε, την, ε, τη σήμανση που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, σε μπούτια κοτόπουλου. Όχι. Το e-labeling, η ηλεκτρονική δηλαδή σήμανση, θα αφορά μόνο προϊόντα, αγαθά, τα οποία έχουν μια ηλεκτρονική οθόνη, μια ψηφιακή οθόνη. Δεν είναι δυνατόν να αφορούν κοτόπουλα. Ε, αυτό δεν είναι προπαγάνδα, είναι στοιχεία. Δεν μιλούμε για σεισμούς, μιλούμε για τεκμηριωμένα στοιχεία. Μετά, πώ θα λειτουργήσουν συμφωνίε και πώ θα ξεπεράσουμε τι δυσκολίε. Ε, ας έχουμε υπόψη μα ότι η ρυθμιστική συνεργασία δεν δημιουργεί μια καινούρια νέα ενιαία αγορά Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτειών. Δεν πρόκειται να δημιουργηθεί καινούριο παράγω που θα κατησχεί της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Πρόκειται απλώς για μια συνεργασία προς την κατεύθυνση των κοινών συμφερόντων όπου υπάρχουν. Αν όμως υπάρχουν διαφορές δεν είναι δυνατόν να συνεργαστούμε. Για παράδειγμα, ε, ε, για τις ε, ορμόνες ή για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Εκεί έχουμε τόσο μεγάλες βασικές διαφορές που δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Όμως υπάρχουν τομείς στους οποίους μπορούμε να πετύχουμε πράγματα, για παράδειγμα την αυτοκινητοβιομηχανία. Εκεί μπορούμε να εξασφαλίσουμε αμοιβαία αναγνώριση των τεχνικών κανονισμών που έχουν αποδειχθεί ότι έχουν παρόμοια ή συγκρίσιμα αποτελέσματα. Αν ένας από τους κανονισμούς προσφέρει μεγαλύτερη προστασία, όπως για παράδειγμα στις ΗΠΑ ε, υπάρχουν κάποιοι κανόνες για τις εκπομπές που είναι πιο αυστηροί από τους δικούς μας, τότε θα ε, επιλέγουμε τον πιο αυστηρό κανονισμό. Σε, στις εκπομπές διοξείδου του άνθρακα όμως οι δικές μας ε, προδιαγραφές είναι πιο αυστηρές, θα εφαρμόζονται οι δικές μας εκεί μπορεί να γίνει ρυθμιστική συνεργασία και να δώσει ωφέλη. Τέλος, <clears throat> μιλάμε για τους ε, δασμούς ε, και για άλλα παραδείγματα. Ας μην υποτιμούμε τους δασμούς. Για παράδειγμα, στην εισαγωγή αυτοκινήτων είναι 10%, στην εφαντουργία είναι 12% και μπορούμε να φτάσουμε και σε δασμούς μέχρι και 30%. Ευτυχώς, τα iPad στις ΗΠΑ είναι πιο φτηνά, όχι εξαιτία των δασμών όμως, ε, έτσι κι αλλιώς όλα τα προϊόντα τεχνολογίας ε, ε, εξαιρούνται της, των δασμών, οπότε υπάρχουν άλλοι λόγοι που εξηγούν τη διαφορά τιμών. Ευτυχώς, για τα iPad. Παρ' όλα αυτά οι δασμοί εξακολουθούν να είναι σημαντικό θέμα, μην το υποτιμούμε. Τέλος, σε ορισμένου τομεί, όπως τα συστήματα τυποποίησης, όπως και την αξιολόγηση συμμόρφωσης, φοβούμε ότι οι προσεγγίσεις από τις δύο μεριές του ωκεανού είναι πολύ διαφορετικές και γι' αυτό λόγο θα πρέπει να εργαστούμε πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ. Thank you. I'm Elena I work Ευχαριστώ, Ελίνα Λόρναν. Θα σε διακόψω όμως, Ελίνα. Θα ξανακούσουμε, ελπίζω, την Επιτροπή. Γιατί μπορούμε να σας έχουμε πότε θέλουμε. Ελπίζω. Αλλά θα πρέπει να ακούσουμε τα σχόλια από τους ε, λοιπούς εμπειρογνώμονες. Καλύτερα. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα εκείνους. Σας υπενθυμίζω. Ότι δεν πρέπει να περιοριστεί ο βαθμός εμπιστοσύνης που έχουμε. Αυτό είναι πάγια απέτηση. Ποιος θέλετε να ξεκινήσει, έχετε κάποια προτίμηση. Ό,τι νομίζετε εσείς. Σημειώνω όμω πάλι ότι και ο Ζάξος είναι πιο εύκολο να έρθει πάλι. Καλώ θα τα ακολουθήσουμε τη σειρά που είχαμε και στην αρχή. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Για το εάν είναι τέλεια η ευρωπαϊκή αγορά για τις ομιθείς. Όχι, προφανώ έχει ατέλειε. Χρειάζεται βελτίωση, το σημειώνουμε. Η αδιαφάνεια κυρίως είναι για μένα πρόβλημα. Και εδώ έχουμε μια διάταξη περί διαφάνειας που καλύπτει όλες τις δημόσιες προμήθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν καλύπτει αντίστοιχα το επίπεδο των ομόσπων των πολιτιών στις ΗΠΑ. Και αν θέλουμε να κοιτάξουμε τι είδου συνέπειε μπορεί να έχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις ως προς τη δυνατότητα για αλλαγή με στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα είναι ένα τομέας μπορώ να απαντήσω. Μπορεί να προσφέρει δηλαδή δυνατότητες για βελτίωση προς το καλύτερο, προς την τελειοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς. Κάτι άλλο... για τις προμηθείες και τις προδιαγραφές επιδόσεων, δηλαδή το επίπεδο της ε, ασφάλειας που επιτυγχάνεται, όχι προδιαγραφές που θα μας οδηγήσουν στον να αγοράσουμε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, προδιαγραφές σχεδιασμού δηλαδή, αλλά προδιαγραφές τις οποίες πρέπει κανείς να τηρεί στο επίπεδο που θέλει μπορεί να τις ορίσει, που όμως δεν μπορούν να αποβαίνουν εις όφελος του ενός προμηθευτή του άλλου. πρόοδος. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε πρόοδο στο επίπεδο των πολιτιών, των ομοσπονδιών πολιτιών. Δεν λέω ότι δεν περιλαμβάνονται οι πολιτείες. 37 πολιτείες καλύπτονται από τις ε, αρχές για τις δημόσιες προμήθειες στις ΗΠΑ, αλλά δεν είναι όλες και δεν είναι όλοι τομείς. Πόλεις ή πολιτείες που καλύπτονται, γιατί καλύπτεται και το Σικάγο ως πόλη, ε, πιέζουμε να ε, προχωρήσουν σε περισσότερη πρόοδο προς την κατεύθυνσή μας και αυτό δεν είναι δύσκολο γιατί ήδη έχουν κάνει κάποιες ε, ρυθμίσεις ικανοποιητικέ. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις όπου έχουμε νομοθετικά όργανα των πολιτιών που αφαιρούν από τον κυβερνήτη που είχε στο παρελθόν τη σχετική εξουσία γιατί θέλουν να διατηρήσουν ως ομοθετικά όργανα την εξουσία πάνω σε αυτές τις προμήθειες. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο για μα. Και γι' αυτό εάν μπορέσει το Κοινοβούλιο σε επαφή με αυτά τα ε, νομοθετικά σώματα, τα τοπικά κοινοβούλια να κάνει κάτι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Μια πολύ δύσκολη ερώτηση για το τι θα πρέπει να παραχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πείσει τις ΗΠΑ. Κοιτάξτε, είναι ζήτημα αμοιβαιότητας. Κάτι θα μας δώσουν, κάτι θα τους δώσουμε. Το θέμα είναι όμως τα αφορά της προμήθειας ειδικά. Οπότε θα πρέπει και η αμερικανική πλευρά να εξασφαλίσει ευρύτερη κάλυψη Φιρυπίν για το επίπεδο των ομοσπονδών κρατηδίων, πολιτιών δηλαδή, ε, δημόσιες υπηρεσίες θα αφορά τοπικές αρχές και κατασκευαστικό κλάδο που ακόμα δεν καλύπτεται. Θα είναι αυτά που θα κάνει, στα οποία θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια παραχώρηση, γιατί αυτά δεν καλύπτονται από τι αμοιβαίε διαπραγματεύσει. Μπορεί να χρειαστεί και να γίνουν παραχωρήσει. Αλλά υπάρχει και το γενικότερο ζήτημα. Παραχωρήσει δηλαδή σε άλλο κεφάλαιο τη TTIP. και αυτό κομμάτι των διαπραγματεύσεων είναι, θα κρυθεί. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η TTIP επειδή αφορά ρυθμιστικά ζητήματα δεν είναι κάτι το οποίο καλύπτει με την σύναψη της απόφασης τα πάντα. Η πραγματική δουλειά γίνεται στην πορεία μέσα από, τις από τα διάφορα σώματα που θα θεσπιστούν ε, για να συνεργαστούν μεταξύ τους. Άρα δεν κρίνεται ε, σε επίπεδο αμοιβαιότητας αυτό αλλά σε επίπεδο ρυθμιστική συνεργασία πολύ περισσότερο από ότι σε μια εμπορική συμφωνία. Όταν έχουμε να κάνουμε δασμού φερρυπίν, ε, ανταλλάσσουμε τον δασμό για ένα προϊόντα σχέση με τον δασμό για ένα άλλο. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε την ίδια κατάσταση όμω, από ό,τι βλέπω εγώ τα πράγματα. Ευχαριστώ Πέτρο και η Ευχαριστώ πολύ. Ε, Καταρχά σα ευχαριστώ για τι ερωτήσει. Πολλέ ήταν και είναι και η μεγαλύτερη μου ανταμοιβή για όλη τη δουλειά που έχω κάνει, το ενδιαφέρον που δείχνετε. Θα ήθελα σύντομα να απαντήσω σε κάποιε ερωτήσει, τέσσερι συνολικά, και ταυτόχρονα να σχολιάσω κάποια από τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Καταρχάς, το, η θεωρία ότι είναι υψηλότερο το επίπεδο προστασία του καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αληθεύει. Έχει αυστηρές ε, προποθέσει, ειδικά αστική ευθύνη, το σύστημα των ΗΠΑ. Και η ενίσχυση του επίπεδου ασφάλειας μέσα από τη ρυθμιστική συνεργασία προκύπτει από τη δυνατότητα να διδαχθεί ο ένας από τις εμπειρίες του άλλου. Για την ερώτηση του κύριου Βουλευτού που αφορά την παρατήρησή μου για τη σχετική σημασία των δασμών. Όντως, σωστά λέτε ότι έχουν σημαντικό ρόλο στην TTIP, σχετικό όμως ρόλο, σχετικό, σχετική σημασία γιατί θα εξαρτηθούν από την θα μπορούν να αναδιαμορφωθούν δηλαδή από τη ρυθμιστική συνεργασία. Για το σχόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Τηλέμα στηρίζεται σε γεγονότα. Ναι, αλλά ξεκινούμε από τις προτάσεις που προκύπτουν στο παρελθόν, από ιστορικές δηλαδή προσπάθειες για τη ρύθμιση των ε, εμπορικών συναλλαγών, αλλά και από το επιστημονικό έργο που έχει μέχρι τώρα γίνει. Γι' αυτό και σας λέω ότι είναι απίθανο να ε, μην επηρεαστεί, να επηρεαστεί διορθώνει η ομιλήτρια το αποφασιστικό, το ρυθμιστικό σύνολο ε, αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά πάλι μια υπόθεση είναι μόνο, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία να υφίσταται και δεν μπορούμε να κάνουμε αξιολόγηση συνεπειών παρά μόνο όταν θα υπάρχει αυτή η διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω στις, ε, στις, στη γραμμή των παρατηρήσεων της Επιτροπής και των εξαιρέτων απαντήσεων της Μπάρμπαρα. Θα ε, βεβαίως σε σχέση με τις πολύ αρθινές ε, και πολύ καλές ερωτήσεις που διατυπώθηκαν και θα απαντήσω και για την ρυθμιστική συνεργασία και γιατί δεν θεωρούμε ότι μπορεί να επηρεαστεί η ρυθμιστική αρμοδιότητα. Νομίζω ότι λάβατε για το πρώτο κομμάτι επαρκείς απαντήσεις. Εάν θέλετε δεδομένα, εάν καταργηθούν όλοι οι δεσμοί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ θα έχουμε 11% αύξηση του ΑΕΠ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 0,11 για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 0,04% για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα το πόσο θα βελτιωθεί η ευημερία μας σχέση με την κατάργηση των δασμών είναι πολύ υπερβολική πρόβλεψη. Από την άλλη βεβαίως αν υπάρξει και πλήρης, θα εξαρτηθεί από το αν θα είναι πλήρη η ρυθμιστική συνεργασία. Θα συνεχίσω στα όσα είπε η Μπάρμπαρα. Στο κείμενο της Επιτροπής με τις προτάσεις ε, προτείνεται δουλειά από ένα ρυθμιστικό ένα, από ένα σώμα ρυθμιστική συνεργασία. Πολλή από τη δουλειά αυτή θα γίνει λοιπόν μετά τη σύναψη τη συμφωνία και οι σχετικέ διατάξει αναφέρονται αντίστοιχα και στην ε, ΣΕΤΑ, στην Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά. Με ενθάρρυνση που αναφέρεται για, τις, ε, για τους εκπροσώπους και τα σώματα των διαφορών εμπορικών δραστηριοτήτων, ε, να συνεργαστούν μεταξύ τους. Υπάρχουν συντονιστές για την απάλληψη των ε, τεχνικών φραγμών κτλ. Ξέρετε δηλαδή από το είδος της δουλειάς που θα θεσπίσουν οι διαπραγματευτές, το είδος της ρυθμιστικής συνεργασίας, τις προτεραιότητες που θα ορίσει ένα έτος, την ποιότητα της δουλειάς συνολικής και αναλόγως θα δούμε ενδεχομένως καλή συνεργασία ή μπορεί και να χρειαστούν κανένα δύο χρόνια μέχρι να δούμε αυτά κάποια κέρδη από αυτή τη συνεργασία. Νομίζω ότι για τη ρυθμιστική αρμοδιότητα καλύπτει η Μπάρμπαρα επαρκώ αυτά που είχα να πω, δηλαδή ότι δεν υπάρχει τελικό κείμενο και σχεδόν δεν μπορούμε να κάνουμε 100% ασφαλεί προβλέψει για το αν θα επηρεαστεί η ρυθμιστική αρμοδιότητα ή όχι. Αυτό που έχω να πω πάντω είναι ότι στο κείμενο των προτάσεων τη Επιτροπή γίνεται μια πρόταση για ρυθμιστική συνεργασία σε σώματα τα οποία όμω δεν θα έχουν αρμοδιότητα για θέσπιση κανόνων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα χάσει από, τα, από τι αρμοδιότητε του μερίδιο. Πάλι δηλαδή θα πρέπει να, περνάει, να περνάει η διαδικασία μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο δε κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπονται και διασφαλιστικοί όροι οι προϋποθέσεις όπου μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επανέρχεται και να παρεμβαίνει στη δικασία αν βλέπει ότι υπάρχουν ζητήματα παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών γενική πολιτική. Άρα και δεν προβλέπεται άμεσα παραβίαση των, ή ε, ε, περιστολή των αρμοδιοτήτων ρυθμιστικών του Κοινοβουλίου και υπάρχει ασφαλιστικη δικλίδα για την ανάκτηση όπου χρειάζεται. Είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι ίσως χρειάζονται περαιτέρω έρευνες στον τομέα αυτό όταν θα είναι έτοιμο το κείμενο και έτσι μπορούμε να σας δώσουμε περισσότερη και πιο ακριβή ανάλυση για τις συνέπειες της ε, ρυθμιστικές Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω δύο ερωτήσεις. Την ερώτηση της κυρίας Γκέμπχαρτ για την ισοδυναμία, για την ισοτιμία θα την απαντήσω ως εξής. Η ισοτιμία έχει χρησιμοποιηθεί προβλέπεται στη συμφωνία TBT στον ΠΟΕ αλλά χρησιμοποιείται ελάχιστα. Υπάρχει μια συμφωνία κτηνιατρική ισοδυναμία του 1998 μεταξύ των ΗΠΑ και τη Ευρώπη, και θα μπορούσε κανεί να πει ότι οι συμφωνίε για τα αεροσκάφη του 2009 και τα ε, βιολογικά πρότυπα πλησιάζουν μια συμφωνία ισοδυναμία. Δεν έχει προσταθεί ε, από όσο ξέρω μέχρι στιγμή κάτι τέτοιο για τα βιομηχανικά προϊόντα αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται στον τομέα, γιατί η έκθεση δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Ισοδυναμία σημαίνει αμοιβαία αναγνώριση, μεν, αλλά λίγο διαφορετική. Και θέλω να σας πω τώρα σε τι ακριβώς συνίσταται αυτή η διαφορά για να καταλάβουμε μια και καλή. Με την ισοδυναμία η χώρα εισαγωγής αποφασίζει κατά πόσο μέσω αμοιβέ αναγνώριση οι εξαγωγέ μπορούν να βασίζονται στου οικείου κανόνε. Ε, ε, η ισοδυναμία είναι πιο περιοριστική. Εάν εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει ισοδυναμία από τη ΣΥΠΑ, αποφασίζει κατά περίπτωση η αμοιβαία αναγνώριση έχει μια αρνητική λίστα αυτή την προσέγγιση ενώ με την ισοδυναμία εξετάζονται οι υποθέσεις ξεχωριστά αλλά υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις οι στόχοι πρέπει να είναι ίσοι, όχι γενικοί στόχοι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι αυτοί οι στόχοι ε, ακριβείς ε, συγκεκριμένοι στόχοι όπω για παράδειγμα στα κτηνιατρικά θέματα, επίσης αποτελεσματικότητα και εμπιστοσύνη και στη κτηνιατρική συμφωνία διατυπώνται πολύ σωστά. Ε, ισοδύναμη επιμέλεια, έτσι αναφέρεται, ίση επιμέλεια. Θα μπορούσε αυτό να ισχύσει και για τα βιομηχανικά προϊόντα. Ε, στο παρελθόν που ανέφερε ο Φερνάντος, ε, προϊόντα ε, τεχνολογίας πληροφορικής. Θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί και στις υπηρεσίες εντός της εσωτερικής αγοράς. Έχουμε κάτι που πλησιάζει αυτό το μοντέλο. Η αμοιβαία αξιολόγηση και η κυρία Κέπχαρ το γνωρίζει πολύ καλά. Είναι ακριβώς αυτό. Η ισοδυναμία λοιπόν είναι κάτι που μπορεί να γίνει, είναι περίπλοκο, αλλά η υποκείμενη ιδέα είναι ότι υπάρχουν ισοδυναμοί στόχοι και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε χωρίς μια ανοιχτή ε, προσέγγιση, αμοιβαία προσέγγιση που μπορούμε να κάνουμε μόνο στην Ευρώπη, ότι θα μπορέσει να σημειωθεί πρόοδο και σε μια ζώσια συμφωνία αυτό θα ήταν απόλυτα αδύνατο. Ακόμα και σε δύσκολου τομές. Είμαι λοιπόν κάπω ενθουσιώδη για αυτή την προσέγγιση. Το δεύτερο, Ιταλό ε, εκπρόσωπο, θα ε, είπε τόσο καθαρά που κατάλαβα τα πάντα τις προτάσεις. Μπορώ να τις, ε, σας τις πω λεπτομερώς. Αλλά κάποια χράματα, ξέρετε, χρειάζονται χρόνο. Χρειάστηκα 20 λεπτά για να, εξηγήσω, για να το εξηγήσω βήμα προς βήμα. Εξηγούνται όλα στο έγγραφο. Και χαίρομαι που η Κομισιόν και όλοι οι εμπειρογνώμονε είπαν ότι η δουλειά που έχει γίνει στο χαρτί είναι σωστή, αλλά χρειάζεται πολλή χρόνο για να παρουσιάσει κανεί όλε αυτέ τι τεχνικέ προτάσει. Και αν δεν μου δώσει η κυρία Φόρντα το χρόνο που χρειάζομαι, θα πρέπει να σας παραπέμψω στο δεύτερο μισό του εγγράφου και στην υποσημείωση που περιέχει όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά υπάρχουν πολλές προτάσεις που θα μπορούσαν να ανοίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ. Δεν είναι λεπτομέρειες προτάσεις για το τι θα μπορούσαν να κάνουν οι οργανισμοί τυποποίησης, αλλά σίγουρα αν συζητηθεί συνεργασία για ένα προϊόν, ε, για ένα πρόγραμμα, θα, θα υπάρξουν προγράμματα στο πλαίσιο της όσας ε, συμφωνίας πολλά είναι δυνατά εφόσον ε, υπάρχει το σωστό πνεύμα στο πλαίσιο της TTIP. Ευχαριστούμε. Θέλω να προλάβετε για τις ερωτήσεις σας, αλλά το επόμενο θέμα της ε, ημερήσιας διαταξής είναι η επέκταση της ψηφιακής αγοράς για τι της ενιαίας αγοράς για την ψηφιακή εποχή και με βέβαια θέλετε να το συζητήσουμε. Οπότε δεν θα ζητήσω περισσότερα τώρα από του εμπειρογνώμονε κομισιών. Θα ζητήσω από τα μέλη να μου πούν κατά πόσο θέλουν να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό σε επόμενη συνάντηση τη Επιτροπή και υποψιάζομαι ότι θα πείτε ναι. Στο μεταξύ, εμεί θα δημοσιεύσουμε όλα αυτά τα έγγραφα, θα σα τα κοινοποιήσουμε, θα σα πούμε πού υπάρχουν ήδη αλλά θα αναφέρουμε στο εξώφυλλα από πού προέρχονται και αν μπορούσατε να μας στείλετε την αναθεώρηση αυτής της, τελικής, της τελευταίας ε, παρουσίασης που κάνατε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο να σας πω η διαπραγματευτική ομάδα της Κομισιόν ε, θα είναι διαθέσιμη για να σας ενημερώνει για οποιασδήποτε εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο ώστε εσείς να παρακολουθείτε τα όσα διαπραγματευόμαστε, το κατά πόσο υπάρχει συνοχή με το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε το Κοινοβούλιο να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο του ως νομοθέτη και ε, ρυθμιστικής αρχής. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να κλείσουμε τη δημόσια συζήτηση γι' αυτό, διότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, απλότητα και γλώσσα που ο κόσμος να μπορεί να καταλάβει. Οπότε θα δώσουμε περισσότερο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ για τις ε, απόψεις και σκέψεις σας. Οτιδήποτε θέλετε, ε, οτιδήποτε μας στείλετε θα το δημοσιεύσουμε. Το επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη είναι μια ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της Επιτροπής ε, από την DG Connect και την DG για την ανακοίνωση της Επιτροπής σε σχέση με τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης. Θέμα που έχουμε συζητήσει ήδη πολλές φορές. Πίτερς. Οι αξιωματούχοι της Κομισιόν για την Τίτη παρακαλούνται να αναχωρήσουν. Όχι, δεν εκτιμάμε την παρουσία σας, την εκτιμάμε, αλλά έχουμε μείνει πίσω χρονικά. Οι ομιλητέ μας είναι ο Ερικ Πίτερς από την DigiConnect. Ο Lionel από την Connect και η Μαρία Χαϊμπάντορ, αρχής από την DG Grow. Peter, θα μας κάνεις μια πρώτη γρήγορη παρουσίαση. Όλοι έχουμε διαβάσει την πρόταση πολλές φορές. Πέντε λεπτά στον καθένα από τους ομιλητές και μετά συζήτηση με τα μέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλύτερα να δώσουμε περισσότερο χρόνο στις ερωταποκρίσεις σήμερα. Θα είμαι λοιπόν πολύ σύντομος. Με συνοδεύουν συνάλφοι της γενική Διεύθυνσης Grow, ε, της γενική Δραματείας και άλλοι για να σας δείξουμε ότι πρόκειται για ένα ομαδικό project. Θα επανέλθω σε αυτό. Ε, ορισμένα στοιχεία, σε ό,τι φορά το περιεχόμενο, να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για προτεραιότητα του Πρόεδρου. Ε, δεν υπάρχουν και πολλές προτεραιότητες, 10, οπότε είναι σημαντικές και οι 10. Είναι μία από τις 10. Η ψηφιακή οικονομία είναι λοιπόν προτεραιότητα της Κομισιόν αλλά αυτό είναι κάτι σχετικά καινούριο. Πριν από πέντε χρόνια δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Οπότε είναι θέμα απόφαση του Προέδρου, αλλά είναι και θέμα εξέλιξη τη κοινωνία και τη οικονομία. Η ψηφιακή στρατηγική επίση ε, συγκεντρώνεται, επικεντρώνεται σε ένα αριθμό μέτρων, 16 μέτρα σε τρει πυλώνε και σε μία περίοδο 18 μηνών. Πρόκειται για, μια ρεαλιστική, για ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, για μια ρεαλιστική πρόταση ε, που ήταν αποτέλεσμα εσωτερικών, μακρόχρονων εσωτερικών διαπραγματεύσεων εντός της Κομισιόν. Το... Μεταξύ των μέτρων δεν υπάρχουν προτεραιότητες, όλα θα πρέπει να εφαρμοστούν στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, 18 μήνες, οι προτάσεις ε, θα υποβληθούν στο τέλος του χρόνου ε, και όλα θα πρέπει να εφαρμοστούν το 2016. Τώρα, έχουμε θέματα όπως τα δικαιώματα του δημιουργού, ε, τα, δικαιώματα, τα, τις συμβάσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου, προστασία καταναλωτών ηλεκτρονικού εμπορίου κλπ. τα οποία ε, είναι λιγότερο τεχνικά. Υπάρχουν όμως και πιο τεχνικά θέματα όπως οι πλατφόρμες, τα δεδομένα κλπ. Τα οποία χρειάζονται περισσότερο χρόνο, πλατφόρμες για παράδειγμα. Ε, εκεί θα πρέπει να γίνει μια σε βάθος αξιολόγηση, οπότε αυτά θα καθυστερήσουν λίγο πιο πολύ από τα προηγούμενα. Αλλά χωρίς να αποτελούν δεύτερη προτεραιότητα. Δεύτερο στοιχείο, χαρακτηριστικό της καινούργιας προσέγγισης κομισιών, είναι, όπως έλεγα και πριν, η ομαδική εργασία. Έχουμε προτεραιότητες στρατηγική μας, ε, οι προτεραιότητες αυτές είναι πολύ όριμες, ε, τις έχει επεξεργαστεί ε, η Κομισιόν, ο πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι, οι επίτροποι που είναι συναρμόδιοι. Όλα αυτά εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, ομαδικής δουλειάς και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ, εκπροσωπούμε διαφορετικές γενικές διευθύνσεις ακριβώς επειδή πρόκειται για μια δουλειά ομάδας. Μάλιστα, συνεργαζόμαστε και με τα κράτη-μέλη και, με και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μένουμε κλεισμένοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε. Ε, μόνο μέσω ενός διαλόγου στην αρχή της διαδικασίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτός ο διάλογος να γίνει στην αρχή πριν υποβληθούν οι προτάσεις. Και ο διάλογος αυτός θα πρέπει να γίνει σε πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά τα επίπεδα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα κλείσω λέγοντας ότι μία από τις προϋποθέσεις για την επιτυχία είναι, θα είναι όλα τα κείμενα τα σχετικά με τη ψηφιακή οικονομία, ε, προστασία προσωπικών δεδομένων, ε, ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, δίκτυα κλπ. Όλες οι προτάσεις οι οποίες τρέχουν αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν έγκαιρα και το αποτέλεσμα να είναι φιλόδοξο όπως είχε εξ αρχής στόχο η Κομισιόν. Αυτά δεν θα πω τίποτα άλλο. Είμαστε στη να απαντήσουμε σε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Κύριος Ζόλα, η κυρία Ριμπάιντερ θα ήθελαν επίσης να παρέμβουν ενδεχομένως. Δεν θέλω να σχολιάσω. Θέλω να συμφωνήσω και να υπογραμμίσω ότι πρόκειται για μια προσπάθεια, πολύ συντονισμένη προσπάθεια πλευράς Κομισιόν. Για την κυβέρνηση Grow ε, έχουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Έχουμε τις ε, πτυχές της εσωτερικής αγοράς αφενός και η ψηφιακή νέα αγορά προφανώς αποτελεί τη της ενιαίας αγοράς και από την άλλη μεριά έχουμε την ψηφιακή οικονομία. Δύο λοιπόν πτυχές διαφορετικές. Δεν θέλω όμως να κάνω κάποια πιο συγκεκριμένα σχόλια προς στιγμή. Κυρία Κέφχαρτ. Θες να κάνεις παρατηρήσεις σου, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμονησύνη μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολήθηκε με τόσο σωτατικό τρόπο με το θέμα αυτό. Καιρός ήταν να αναπτύξουμε μια στρατηγική για το πώς θέλουμε να χειριστούμε τους τομείς αυτούς. Θα υπενθυμίσω ότι και από και εμείς στην Επιτροπή μας έχουμε από το 2011 μια ομάδα εργασίας η οποία ασχολείται με τα θέματα αυτά. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε μια σειρά από πράγματα, πολύ σημαντικό, κατά με. Πρέπει πολύ γρήγορα να τα διευθετήσουμε. Χαίρομαι που συμφωνεί σε αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα στον τομέα του εμπορίου μέσω του διαδικτύου, το e-commerce εν γέννη. Διαπιστώνουμε δηλαδή εκεί ότι παραμένουν πολλά προβλήματα, πολλές δυσκολίες για τις επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες κυρίως, προβλήματα που πρέπει να ξεπεράσουμε, αλλά και για τους καταναλωτές. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε και να βρούμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις και γι' αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερως για το ότι όπου υπάρχει ανάγκη για ρυθμίσει, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως θα είναι έτοιμη στο τέλος του χρόνου να θεσπίσει διατάξεις στο θέμα του ενοχικού δικαίου και με έναν τρόπο που θα εναρμονίσει τους κανόνες. Δηλαδή έχουμε πλέον αλλαγή ρότα σε σχέση με την προηγούμενη επιτροπή που είχε ένα σύστημα. σύστημα. Αυτό είναι καλό και για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και για τον καταναλωτή. Πολύ καλή εξέλιξη. Μια ερώτηση την οποία έχω πάντοτε διατυπώσει και την επαναλαμβάνω εδώ όταν μιλούμε για το geo-blocking. Γίνεται λόγος για μη θεμητό geo-blocking, το οποίο πρέπει να καταργηθεί, να απαγορευτεί. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό τι σημαίνει αθέμητο και ποιο είναι ενδεχομένω το δικαιολογημένο ή θεμητό geo-blocking. Δεν μου έχει δώσει κανείς ακόμα απάντηση. Μήπως τα καταφέρουμε σήμερα. Τρίτη ερώτηση. Για το κατά πόσον έχει η Επιτροπή ενασχοληθεί με το πρόβλημα των αποκλήσεων μεταξύ των διατάξεων που αφορούν το online και το offline, των, τις συνοριακές και τις μη συνοριακές αγορές αγοραπολισίες. Θα ήθελα λοιπόν να αποφύγουμε τον κίνδυνο αυτό, γιατί θα ήταν κακό και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τον καταναλωτή να υπάρχει τόσος κατακαιρματισμός διατάξεις. Και γι' αυτό ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι είδους προσέγγιση μπορεί να υιοθετήσει για να δώσει λύσεις. Και άλλη μια παρατήρηση, ε, η ερώτηση, αν και θα είχα πολλές περισσότερες, στις εξελίξεις στην ψηφιακή εσωτερική αγορά, βλέπω ότι τα όρια μεταξύ υπηρεσιών, παρόχων υπηρεσιών και προϊόντων γίνονται όλο και πιο ασαφή. Παλιότερα μπορούσαμε να πούμε, να αυτό είναι ένα προϊόν και άρα επάγεται στον εξή κλάδο του δικαίου. Ενώ εδώ έχουμε μία υπηρεσία και άρα επάγεται σε άλλο κλάδο δικαίου. Χάνονται σιγά σιγά αυτές οι δυνατότητες διάκρισης ε, ως προς την παροχή των υπηρεσιών. Ο εκτυπωτής, ο τρισδιάστατος Φερρυπίν ή η παροχή υπηρεσίας που ταυτόχρονα μπορεί να προσφέρει και προϊόν και άρα εκεί τίθενται ζητήματα ασφάλειας προϊόντων ή ασφαλούς προϊόντος ή ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ συγκεκριμένα πλέον τα όρια και άρα θα πρέπει να βρούμε τι ισχύει για να έχουμε και την απαραίτητη ασφάλεια δικαίου. Άντε και θα κάνω και άλλη μια ερώτηση γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ που αφορά τη διάκριση και είναι και σχετική με άλλες ερωτήσεις μου προηγουμένως διάκριση μεταξύ του, των διαγραμμικών και μη διαγραμμικών αγοραπολισιών, offline και online. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αυτών ειδών αγοραπολισιών και δεν νομίζω ότι ρόλος του νομοθέτη είναι να υποστηρίξει τη μία ή την άλλη εκδοχή της αγοραπολισίας. Πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα είναι θεμητός ανταγωνισμός που θα αναπτύσσεται. Αυτό είναι όλο. Πώς λοιπόν μπορούμε να καλύψουμε και την ανάγκη να είναι δεσμευτικά, ε, δεσμευτικές νομικά διατάξεις είτε για το online είτε για το offline. Υπάρχουν επίσης ε, πολλές περιπτώσεις όπου μπορεί μια επιχείρηση να πωλεί online αλλά να λέει για την παράδοση του προϊόντος θα περάσετε στο κατάστημα. Αυτό σε, που, σε ποια κατηγορία θα ταξιδονομήσουμε, σε online ή σε offline. Όπως είπα, είναι πολύ ασαφή τα όρια πλέον. Και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε λύσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν μια δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των διαφορών ειδών Merci, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Ε, βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο μιας ε, μακράς μάλλον διαδικασίας ορίμανσης. Η δημιουργία μιας ψηφιακής ε, οικονομίας δεν είναι κάτι καινούριο, πρόκειται για μια μετατροπή της παραδοσιακής οικονομίας σε ψηφιακή οικονομία. Οπότε μην κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι δημιουργούμε, οικοδομούμε κάτι τελείως καινούριο, διότι η παραδοσιακή παλιά οικονομία θα συνεχίσει να υπάρχει και θα μετατρέπεται σιγά σιγά σε ψηφιακή οικονομία. Η Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων ασχολείται με την, ε, και με την καινούρια ψηφιακή οικονομία και με την παλιότερη οικονομία που θα γίνει ψηφιακή. Τώρα, ερώτηση. Σας για το θέμα των δικαιωμάτων του δημιουργού. Γνωρίζουμε τα επιχειρήματα σε ό,τι αφορά την ισορροπία ανάμεσα στην πρόσβαση και την προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού. Ε, πρόκειται για συγκρούσεις αντιφάσεις που ε, θα πρέπει να επιληθούν. Εν πάση περιπτώσει για μένα δεν υπάρχουν καν αντιφάσει. Ε, το... Θέλω να σχολιάσω την γενικότερη ουσία του κειμένου. Πολύ συχνά το κείμενο αναφέρεται στις επιθυμίες της ε, Κομισιόν ε, με έναν τρόπο που δείχνει να βλάπτει τα δικαιώματα του δημιουργού. Για παράδειγμα, ο, ο, τίτλος λέει «Βελτίωση της πρόσβασης σε ψηφιακό δεδομένο, στα ψηφιακά δεδομένα». Ε, εξυγχρονισμός του πλαισίου ε, των δικαιωμάτων του δημιουργού. Όλοι συμφωνούμε με τον εξυγχρονισμό των, του πλαισίου. Έτσι κι αλλιώς γενικώς οποιοδήποτε εξυγχρονισμός είναι καλό στη ζωή. Αυτό όμως δεν αρκεί. Ε, ε, τι κρύβεται πίσω από τον εξυγχρονισμό. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα. Επίσης άλλες φράσεις που λέει θα, ίσως θα, θα είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η νομική ασφάλεια έτσι ώστε να επιτρέψουμε τους ε, ερευνητές, να, ε, στους ε, ερευνητές, στους αναζητώντες για την ακρίβεια, να έχουν πρόσβαση σε υλικό το οποίο προστατεύεται από το δικαιώμα του δημιουργού. Μου φαίνεται ότι η γενικότερη φιλοσοφία του κειμένου αμφισβητεί την παραδοσιακή έννοια του δικαιώματο του δημιουργού. Οπότε αυτή είναι μια γενική μου Σε ό,τι αφορά την, τοπική εφαρμογή ε, άσκηση των δικαιωμάτων του δημιουργού ε, μερικές ε, φορές οι περιορισμοί αφορούν πιο πολύ εμπορικά δικαιώματα και όχι δικαιώματα του δημιουργού δηλαδή κάποιοι οποίοι έχουν κάποια εμπορικά δικαιώματα επί ενός προϊόντος αποφασίζουν να μην τον διανύμουν ή να μην τον εμπορευτούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή εξαιτίας του ότι το κόστος ε, θα ήταν μεγαλύτερο από το κέρδος. Συνεπώς, ε, σε τέτοιες περιπτώσεις τα δικαιώματα του δημιουργού δεν εμπλέκονται καθόλου. Θα ήθελα να μου πείτε και για αυτό το θέμα ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά την ε, τοπική χρήση ή τον τοπικό περιορισμό της άσκησης των δικαιωμάτων του δημιουργού ε, δεν θα πρέπει να αμφισβητήσουμε ε, ισορροπίες οι οποίες έδωσαν στην ε, Ευρώπη τον χαρακτήρα μιας ε, δημιουργικής περιοχής. Η Ευρώπη είναι μια περιοχή δημιουργίας ε, και η δημιουργία θα πρέπει να προστατεύεται. Γιατί αν δεν προστατέψουμε την δημιουργικότητά μας θα πάψουμε να είμαστε οτιδήποτε. Δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε την προσέγγιση των μεγάλων οικονομικών παραγόντων που βλέπουν τη, τα, μόνο σε εμπόρευμα τη δημιουργία αυτή. Ευχαριστώ, θα μιλήσω ο, εκ μέρους του ECR και θα είμαι κι εγώ σύντομη όσο μπορώ. Καταρχήν, όταν ομοθετούμε σε αυτό το σημαντικό τομέα θα πρέπει να εξασφαλίζουμε, να διασφαλίζουμε ότι ε, στηρίζουμε τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής επανάστασης και όχι ότι θα την υποσκάπτουμε. Θα πρέπει να ε, οι προτάσει μας να είναι τεχνολογικά ουδέτερες, να ξέρουμε ότι η ψηφιακή αγορά είναι παγκόσμια αγορά, όχι ε, όπως οι κάποιες άλλες παραδοσιακές παλιότερες αγορές, μη ψηφιακές, και επίσης θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τον αντίκτυπο που θα, έχουν, θα έχει η καινούργια μας νομοθεσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ε, μικρές επιχειρήσεις και την καινοτομία. Η στρατηγική της Κομισιόν έχει καλά στοιχεία αλλά μπορεί να βελτιωθεί, κατά την άποψή μου, και η Επιτροπή μας θα πρέπει να κάνει αυτό που κάνει πάντοτε καλύτερα, δηλαδή να εστιάσουμε σε πρακτικές λύσεις έτσι ώστε να μειώσουμε τα εμπόδια στο εμπόριο, βοηθώντας και τις επιχείρησεις και τους καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του καταναλωτή, θα ήθελα να ενθαρρύνω ε, ω και ο από την την Κομισιόν, να συγκεντρώσει τις προσπάθειές σας, τις προσπάθειές να, να, εστιάσει και να γίνει πιο συγκεκριμένη. Ε, για δύο χρόνια ζητούσαμε το θέμα των ε, δικαιωμάτων τελικού χρήστη ε, και αυτό που ζητούσαμε ήταν ε, αν ο πάρχος του ίντερνετ δεν σας δίνει την ταχύτητα που έχει υποσχεθεί, την ποιότητα γενικότερα που ε, είχε υποσχεθεί να μπορείτε να ξαναδιαπραγματευτείτε το, ε, τη σύμβαση ή να την ακυρώσετε. Μόνο αυτό ζητάμε και ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει στον τριμερή διάλογο. Οπότε παρακαλώ πολύ να είστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι γιατί προσπαθώντας να λύσουμε όλα τα ζητήματα με μία πρόταση ε, διαμιάς ε, θα αποτύχουμε. Ας είστε λοιπόν πολύ συγκεκριμένοι ποια είναι τα δικαιώματα. Ε, αν δεν μπορείτε για παράδειγμα το, να κατεβάσετε το ψηφιακό δεδομένο, ε, το, τα ψηφιακά δεδομένα που σας έχουν υποσχεθεί, μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο ή κάτι, τέτοιου είδους πρακτικές λύσεις, πρακτικά πράγματα, πολύ συγκεκριμένα θέλουμε από εσά. Και το ίδιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κι εμείς. Σε ό,τι αφορά την επίδοση δεμάτων, ε, είναι πρόβλημα κάπου, όχι παντού. Ε, εμείς ε, έχουμε ε, ορισμένες αγορές που λειτουργούν σωστά. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η διαφάνεια σε όλα τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά το geo-blocking, ε, το δημιουργικό περιεχόμενο είναι από τα ατού Θα πρέπει λοιπόν να το προστατεύουμε, να αρνηθούμε και να καταπολεμήσουμε την πειρατεία, ε, εμείς δεν υποστηρίζουμε πανευρωπαϊκές άδειες, αλλά υπάρχουν τρόπος να στηριχθούν τα δικαιώματα του δημιουργού και να ε, εφαρμόζονται οι κανόνες που υπάρχουν. Ε, να δούμε τους κανόνες ΦΠΑ και το πώς επηρεάζουν τις μικρές επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι κλειδί για την ψηφιακή επανάσταση και επιγόντως θα πρέπει να εξετάσουμε την γραφειοκρατία την οποία θα μπορούσε να εισάγει μια πανευρωπαϊκή άδεια. Για τις πλατφόρμες εξελίσσονται εξαιρετικά γρήγορα σε πάρα πολλούς τομείς. Οι πλατφόρμες στην διαμερασμένη οικονομία αυξάνονται και γιατί τις χρησιμοποιούν οι καταναλωτές. Οπότε έχουν τα πλεονεκτήματα, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα εξασφαλιστεί και ο ανταγωνισμός και η ασφάλεια. Επίσης, θα ήθελα περισσότερα πράγματα για την ασφάλεια ε, στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους ανήλικους. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει το θέμα αυτό να περιλαμβάνεται μόνο στο κεφάλαιο για τις πλατφόρμες. Σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων, οι συνάλφοι της Επιτροπής Λίμπε Πολιτικών Ελευθεριών εργάζονται πολύ προσεκτικά ε, για αυτό το θέμα. Παρακαλώ πολύ έχετε υπόψη σας ότι ε, οι περισσότερε ευρωπαϊκέ επιχειρήσεις είναι B2B, business to business, από επιχείρηση σε επιχείρηση δηλαδή προσφέρουν υπηρεσίε και όχι ε, από επιχείρηση σε καταναλωτές B2C. Οπότε από πλευρά του καταναλωτή, καταναλωτέ ε, δεν θα δούμε με καλό μάτι ε, οι κανόνες προστασία να τους επιβάλλουν τελικά να ανακοινώνουν περισσότερα στοιχεία, να κοινοποιούν περισσότερα στοιχεία. Επίσης είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τα πρότυπα, της προδιαγραφές, ε, ε, να, ε, αυτά να αποφασιστούν από κάτω προς τα πάνω. Ο ψηφιακός κόσμος καινοτομεί πολύ γρήγορα, οπότε θα πρέπει να έχουμε μια συμμετοχική διαφανή διαδικασία στην οποία να μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφέρομενοι και εμπλεκόμενοι φορείς όταν πρόκειται να δημιουργηθεί κάποιο καινούριο πρότυπο Κάτι καινούριο στάνταρ. Αυτά είναι μέσα από τις, αυτές είναι μέσα από τις παρατηρήσεις μας. Ε, θα το ξανασυζητήσουμε προφανώς το θέμα αυτό. Thank you. Κυρία Κάλλας. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είμαι εισηγήτρια και στην Μήτρε. Και ακόμα δεν έχει κλείσει το ζήτημα, ίσως θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε οι δύο επιτροπές μας. Άλλωστε πολλοί και από τους συναδέλφους εδώ είναι μέλη και της Ήτρε. Κάποια αρχικά σχόλια. Νομίζω η οικοδόμηση εμπιστοσύνη είναι το κύριο ζήτημα και ο πυλώνας της στρατηγικής αυτής και ισχύει για τον καταναλωτή όπως και για τις επιχειρήσεις. Συχνά οι επιχειρήσεις δεν αισθάνονται ε, εμπιστοσύνη να πωλήσουν ε, διαγραμμικά γιατί δεν ξέρουν τι είδους διατάξεις μπορεί να ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος για την προστασία του καταναλωτή ή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το καθεξής. Βεβαίως μπορούμε να ισχυριστούμε ότι επιδιώκουμε τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές και προστασία. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε τους ίδιους κανόνες και τις προδιαγραφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση παντού, ώστε ο καταναλωτής να ξέρει τι αγοράζει και με ποιου όρου και το ίδιο και η επιχείρηση να ξέρει τι πολύ και με ποιου όρου. και τι ισχύουν ήδη οι κανόνε εν γέννη. Σημαντικό είναι επίση η Επιτροπή να αντιληφθεί ότι πρέπει να διερευνάτε εάν χρειάζεται να ε, εισαχθεί νέα νομοθεσία για να λειτουργήσει ένα σύστημα ή αν απλώς χρειάζεται καλύτερη υλοποίηση τη φυστάμενης. Ε, παραδείγματι στις, ε, στην οδηγία για τις υπηρεσίες άρχισε τώρα να ασχολείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αποδάθρωση τελικών φραγμών στην ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών και αστεί από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τι σχετικέ διατάξει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να ξεκινήσει αυτή η στρατηγική τη g Market να εφαρμόζεται. Και τελευταίο σχόλιο για τον κύριο Ζουβά. Τι σημαίνει εξυγχρονισμός των δικαιωμάτων του παραγωγού. Ε, αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι το υφιστάμενο δίκαιο δεν έχει λάβει υπόψη του τις τεχνολογικές εξελίξεις. Κάθε στιγμή, κάθε φορά δηλαδή που ε, διαβάζουμε κάτι ή ακούμε κάτι, βλέπουμε κάτι στο διαδίκτυο, το, ο υπολογιστής μας διατηρεί ένα αντίγραφο και περισσότερα μάλιστα αντίγραφα του αρχείου που είδαμε δεν λαμβάνει υπόψη απλώ η νομοθεσία τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τεχνολογία. Αυτό ήταν ένα μικρό σχόλιο για την κυρία Σβέα και πολύ ευχαριστώ να συνεργαστώ μέσα στο εγχείρημα αυτό. Οι πρόεδρο, μπορούν να μας δώσουν διερμηνήσει ακόμη 10 λεπτά και σα ευχαριστούμε. Χωρί αυτό βέβαια να σημαίνει ότι πρέπει να μαγρηγορούμε, πρέπει να είμαστε δυνατόν πιο σύντομοι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρέντα, ένα Πράγμα που προέκυψε έκυψε όταν ήμουν εισηγήτρια στην αναθεώρηση της οδηγίας ΕΚΟΣΟΚ ε, για το πώς πρέπει να λειτουργεί μια ενιαία ψηφιακή αγορά σε θέματα copyright. Αυτό που προέκυψε από την ψηφοφορία και προέρχεται ουσιαστικά από αυτήν εδώ την Επιτροπή είναι ότι σε μια ενιαία ψηφιακή αγορά ε, για να, η νομοθεσία περί copyright χρειάζεται ένα σαφέ σύνολο δικαιωμάτων των καταναλωτών. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη στρατηγική ενιαία ψηφική αγορά. Δεν συζητάμε λοιπόν απλά περιμείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις. Συζητάμε για τη βελτίωση της κατάστασης για όλους τους χρήστες δημιουργικού περιεχομένου και online υπηρεσιών. Υπό το ίδιο πνεύμα θα ήθελα να ενθαρρύνω την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ευρεία έννοια της έννοιας ψηφιακής αγοράς ως βάση. Μια λέξη που ακούμε είναι ψηφιακή ένωση, ακούγεται αρκετά, όχι απλά εμπορικές συναλλαγές υπό τη στενή έννοια. Η στρατηγική λοιπόν αυτή και όταν συζητάμε για γραφικό αποκλεισμό, για geoblocking, ε, αναφερόμαστε σε πρόσβαση σε συγκεκριμένο νομικά προστατευόμενο περιεχόμενο. Και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα πολλοί κόσμος. Ε, δεν μπορεί, δεν έχει πρόσβαση σε κάποιο περιεχόμενο νόμιμα, διότι απαγορεύεται η πρόσβασή του σε συγκεκριμένε χώρε. Οπότε τίθεται το ζήτημα τη διασυνοριακή πρόσβαση όχι μόνο σε ε, προϊόν που υπάρχει προ αγορά, αλλά και κάτι ενδεχομένω που έχει ε, χρηματοδοτηθεί ε, κρατικά, μέσω κρατικών σταθμών ή και άλλες υπηρεσίε Εκεί αντιμετωπίζει τα προβλήματα γεωγραφικού αποκλεισμού ο μέσος καταναλωτής. Η πολιτιστική ποικιλομορφία εξαρτάται στην Ευρώπη δεν περιορίζεται στα εθνικά σύνορα. Ε, έχουμε πολλούς πολιτισμούς νοοτροπίες που δεν γνωρίζουν συγκεκριμένα σύνορα οπότε οι μειονότητες ορισμένων για παράδειγμα μειονότητες ορισμένων χωρών ε, έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που βρίσκονται στη γλώσσα τους ανεξάρτητα από το αν είχαν την ευκαιρία να τις ε, πληρώσουν ή όχι οπότε δεν πρέπει να είμαστε στενόμυαλοι και να εξετάζουμε μόνο τις εμπορικές συναλλαγές στο πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, όχι μόνο δηλαδή να συζητάμε για πράγματα που ε, παρέχει τη δυνατότητα να αγοραστούν. Στον, όσον αφορά τις πλατφόρμες θα θέλαμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις αλλά υπάρχει και κάποια αντίφαση σε σχέση με τα όσα λέει η στρατηγική τη ενία ψηφιακή αγορά. Έχουμε κάποιε αντιφατικέ ενίε. Από τη μία λέμε ότι οι πλατφόρμες πρέπει να είναι πιο ουδέτερε και από την άλλη πιο ουδε... υπεύθυνε, πιο αξιόπιστε. Αυτό αποτελεί αντίφαση. Από τη μία ουδετερότητα έχουμε αυτή την αρχή που λέει ότι όλε οι δραστηριότητε τρίτων μερών αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Πολύ σημαντική έννοια, αλλά ταυτόχρονα εισάγουμε την έννοια της ευθύνης, της λογοδοσίας, δημιουργώντας δηλαδή κίνητρα ε, για τις εταιρείε να αστυνομεύουν το περιεχόμενο τους και να διαφοροποιούν τη χρήση των πλατφόρμων αυτών. Αυτό πρέπει λοιπόν να το διερευνήσουμε λίγο περισσότερο, να το εξετάσουμε περαιτέρω κατά τη συζήτηση σε αυτή την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σούλη. Αυτή ήταν η ομιλητή για κάθε ομάδα έχουμε την κυρία Άννα Μαρία Κορατσαμπίλτ, Γκουτιέρες Πιέτο, Βάσιντον και Ντάλτον. I will be very brief because of... Uh, Θα είμαι σύντομη. Καλωσορίζω την πρόταση της Επιτροπής. Είχε έρθει πια η ώρα για να περάσουμε σε μια συγκεκριμένη πρόταση και εδώ έχουμε την ευθύνη να προχωρήσουμε γρήγορα κάτι βασικό. Πιστεύω η πρόταση πρέπει να αποσκοπεί σε καθολικό δωρεάν και ελεύθερο διαδίκτυο. Μιλάμε για ψηφιακή εθνική κυριαρχία, ευρωπαϊκό υπολογιστικό νέφος. Πράγματα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη. Το ζήτημα είναι οι επιχειρήσει μας να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, να παρέχουν ε, να παράσχουμε ε, συνθήκες ίσου ανταγωνισμού απομακρύνοντα τα εμπόδια. Το θέμα δεν είναι να κρατήσουμε έξω τι εταιρείε τρίτων χωρών. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε και χαίρομαι που η Κομισιόν ε, σκέφτεται προ αυτή την κατεύθυνση χωρί να πέφτει στην παγίδα κατακρεματισμού του διαδικτύου. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω για σήμερα απλά είναι ότι χαίρομαι που η Κομισιόν εστιάζεται στο ζήτημα του κατακρεματισμού. Η πρόκληση είναι η εναρμόνιση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, η άρση όλων των επιπλοκών και κανόνων που δυσκολεύουν τη δουλειά. Εγώ επειδή είχα μια επιχείρηση διαδικτυακή μπορώ να σας πω εμπειρίες ότι το κατακρεματισμός των διαφόρων καθεστώτων ΦΠΑ και τα προβλήματα στις παραδόσεις το γεγονό ότι έχουμε μεγάλες διαφορές όσον αφορά τα κόστη μεταφοράς και παράδοσης ε, μεταξύ κρατών μελών ακόμα και όταν οι αποστάσεις δεν είναι τόσο μεγάλες αυτό αποτελεί τεράστιο κόστος για μικρές επιχειρήσεις ευχαριστώ Ο κ. όταν μιλάμε για την ψηφιακή οικονομία ε, δεν ε, σημαίνει αυτό ότι κάποιοι καινούργοι κλάδοι θα ε, διώξουν ε, κάποιους παλιότερους παραδοσιακούς. Το αντίθετο, κάποιοι παραδοσιακοί τομείς θα γίνουν ψηφιακοί και αυτό συζητάμε. Η στρατηγική αυτή είναι καλή, είναι ε, φιλόδοξη. Βέβαια τα πράγματα εξελίσσονται και αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα από ότι οι δικές μας στρατηγικές. Ε, και η αναλογική μας οικονομία θα πρέπει πολύ γρήγορα να προσαρμοστεί στην ψηφιακή εποχή και κάποιοι κλάδοι μένουν ε, απ' έξω. Ε, και δυστυχώς χάνουμε χρόνο διότι δεν επωφελούμαστε των μηχανισμών που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι και αυτοκριτική προκειμένου να αποφύγουμε την αύξηση της ανεργίας, ιδιαίτερα σε ορισμένους κλάδους και σε ορισμένες περιοχές, προσαρμοζόμενοι στην καινούργια ψηφιακή τεχνολογία. Η στρατηγική είναι θετική, είναι ε, φιλόδοξη, αλλά έχουμε και άλλους μηχανισμούς. Για παράδειγμα, η κατά χώρα συστάσεις, ε, ξεχρονισμός του καθεστώτος ΦΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο. Δηλαδή μέσω των αναχώρων συστάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμηνού θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια πιο εναρμονισμένη, ένα πιο εναρμονισμένο πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υποφεληθούμε αυτών των ευκαιριών, αυτών των μηχανισμών. Έχουμε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωση που χτίζεται σιγά σιγά με τις πλατφόρμες, με την έλξη των και νέων επενδυτών, με τη δημιουργία πλαισίου, με την αποφυγή δεσπόσας θέσης, ε, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε απαιτητικοί και με τα κράτη-μέλη. Γιατί και αυτά έχουν υποχρεώσεις και είναι απογοητευτικό που η Κομισιόν ακόμα πιέζει τα κράτη-μέλη να κάνουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Για παράδειγμα, εναρμόνιση ΦΠΑ, προσαρμογή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία, κόστη, ε, πλατφόρμες ε, ε, διακίνησης εμπορευμάτων και αγαθών κλπ. Που έχουν σχέση με εθνικές πολιτικές βέβαια. Thank you very much, uh, Κυρία Τούνουν Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκε για το ΦΠΑ. Νομίζω όμω ότι αυτό αναφέρεται σαφώ στην στρατηγική. Λέει η στρατηγική ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με του διαφορετικού συντελεστέ ΦΠΑ και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται εναρμόνιση. Επίση για το θέμα τη επίδοση δεμάτων. Υπάρχει μια πολύ σύντομη και γενική φράση στρατηγική. Σε ορισμένε χώρε το σύστημα λειτουργεί, σε ορισμένε όχι. Αλλά έχουμε και μια ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και γι' αυτόν τον λόγο το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί παντού. Στι 2 η ώρα, σήμερα, γίνεται μια εκδήλωση σε, ένα, σε μια από τι αίθουσε μελών ακριβώ για αυτό το θέμα. Και αν θέλετε, αν σα ενδιαφέρει, ελάτε. Οι ταχυδρομικέ υπηρεσίε σήμερα δεν φαίνεται να ε, υλοποιούν, να πραγματοποιούν τις επιθυμίες των καταναλωτών. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επίδοση θεμάτων. Θα πρέπει ταχύτατα να αλλάξουμε το σύστημα για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Αλλά και για να χρησιμοποιήσουμε και τις δυνατότητες που μας δίνει η ψηφιακή εποχή. Η ερώτησή μου είναι, Υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Υπάρχει κάποιο πιο συγκεκριμένο σχέδιο, κάποια σχέδια από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ε, ενδυναμώσει, να στηρίξει την καινοτομία σε αυτό το τομέα. Χρειάζεται να ε, πετύχουμε μια αλλαγή σίγουρα. Τελευταίο ομιλητής ο Ντάν. Ε, δεν περιμένω Κομισιόν να απαντήσετε τι ερωτήσει σήμερα. Πάρτε τες μαζί σας στο γραφείο σας, σκεφτείτε τες και θα ξαναβρεθούμε από κοντά να μας απαντήσετε. Ακούστε απλώς τα σχόλια και ενδεχομένως μπορείτε να έρθετε και διμερώς σε επαφή με τα μέλη. Ντάν. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όλο και περισσότερο ανησυχώ διαβάζοντα τι προτάσει τη Επιτροπή, γιατί βλέπω να είναι μια παλιά προσέγγιση αυτή που, έχει, υποκαλύτερα να αντιμετωπίσει νέε προκλήσει προστατευτική, προστασία εφιστάμενων ε, ελίτ και κατεστημένων. Μια τέτοια προσέγγιση βλέπω να παίρνει η Επιτροπή, τελείως διαφορετική από αυτό το οποίο προσφέρει στον καταναλωτή η ψηφιακή αρένα. Αυτό μάλιστα σαν επίκριση δεν απευθύνω μόνο στην Επιτροπή αλλά και στο Κοινοβούλιο γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα συζητήσαμε στην Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων για μια απαγόρευση για λήψη φωτογραφιών από τους ανώτερους ορόφους του πύργου Άιφελ, η οποία φαίνεται ότι επεκτάθηκε σε όλα τα υψηλά κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε το ψηφιακό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλο τρόπο. Ε, είναι πολύ δύσκολη πρόσβαση στην αγορά, πρέπει να διευκολυνθεί αυτό, να προσαρμοστούμε στα νέα επιχειρησιακά μοντέλα να μην επιδιώκουμε κανόνες και κυρίως όσον αφορά τις υπηρεσίες που ισχύουν για offline αγορές ε, να τους επιβάλλουμε στην ε, αγοραπολισία online γιατί εδώ ο άνθρωπος θα ψηφίσει πάντα με βάση το πορτοφόλι του. Πρέπει να βρούμε ένα πιο παλόμενο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του αύριο και για το geo-blocking, που βλέπω ότι είναι πολύ περιορισμένε οι φιλοδοξίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται το geo-blocking. Αλλά από την άλλη δεν θέλω και πανευρωπαϊκέ άδειε. Η Επιτροπή φαίνεται να μα λέει το αντίθετο ακριβώ. Ότι θέλει πανευρωπαϊκέ άδειε, αλλά δεν θέλει ε, να υπάρχουν περιορισμοί στο geo εκεί που μπορεί να είναι υποφελή για το οπτικοακουστικό υλικό και ούτω καθεξής. Δεν μα λέτε λοιπόν ε, αν μπορείτε να αλλάξετε και να κοιτάξετε με πιο μοντέρνο τρόπο τα πράγματα. Η κυρία Γκέπχαρτ έχει το λόγο. Μια φράση μόνο. Θέλω να παρακαλέσω στη συζήτηση αυτή που γίνεται εδώ και ειδικά για το geo-blocking. Να μην κοιτάμε το θέμα αυτό μόνο από την οπτική των οπτικοακουστικών μέσων και του πολιτισμού. Υπάρχει και το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν πρέπει να λησμονούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη δική μα Επιτροπή. Πολλοί από του συνάδελφου που τοποθετήθηκαν τοποθετήθηκαν σαν να πρόκειται μόνο για ψηφιακό περιεχόμενο. Όχι, είναι πολύ ευρύτερο το ζήτημα. Δεν μπορούμε να το περιορίζουμε έτσι. Η Πρόεδρο. Ευχαριστώ θερμά. Όπω είπα, δεν μπορώ να κρατήσω περισσότερο του ερμηνεί. Θα έχουμε την ευκαιρία άλλη φορά. Χαίρετε.